Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς έχουμε μια τροποποίηση στη μερίσια διάταξη. Μετά από αίτημα του κυρίου Ταραμπέλα, σας προτείνω να μεταθέσουμε την ψηφοφορία για το Ταμείο Ενίσχυσης των Απόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Επίσης πληροφορώ ότι η κυρία Σάρμπου δεν είναι σε θέση να έρθει στην συνεδρίαση την αυριανή μας. Επομένως σας προτείνω να μεταθέσουμε την ψηφοφορία και για τη δική της την προκειμένου να ψηφίσουμε συνολικά στις 25 Μαρτίου του 2013 για αυτές τις δύο εκθέσεις. Επομένως, η αυριανή συνεδρία θα ξεκινήσει στις 11, ενώ των συντονιστών στις 10. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με αυτές τις τροποποίησεις. Η συνήθιση διαδικασία όσον αφορά τα πρακτικά, δίνω ευθύ αμέσω το λόγο και καλωσορίζω ολόθερμα τον Επίτροπο Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίο είναι αρμόδιο για ζητήματα υπηρεσιών και εσωτερική αγορά, και ο οποίο θα μα μιλήσει για ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την κοινοβουλευτική μα επιτροπή. Θα μα μιλήσει για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε βασικά γεωργικά προϊόντα, καθώ επίση και για τις συμπεράσματά του όσον αφορά το φόρουμ υψηλού επίπεδου για μια καλύτερη λειτουργία τη τροφική αλυσίδα. Θα μα μιλήσει επίση και για του στόχου του στα πλαίσια τη πράσινη βίβλου όσον αφορά τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ. Αγαπητέ Μισελ, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στην Επιτροπή μας. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο γιατί ξέρω ότι πρέπει να φύγετε στις 4 εξαιτίας της κρίσης στην Κύπρο. Ζητώ λοιπόν ευθύ αμέσω από του συναδέλφου να μα πούνε ποιοι θέλουν να πάρουν το λόγο αμέσω μετά για ερωτήσει ή παρατηρήσει. Αγαπητέ Μισελ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πάολο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρίσκομαι εδώ με τον πρόεδρο με τον οποίο ως ε, πρώην Υπουργό Γεωργίας πριν απο τρια τρία-τεσσέρα χρόνια συνεργαστήκαμε πάρα πολύ, θα ήθελα να σας ε, χαιρετήσω όλους εσάς τους παρόντες στην Επιτροπή αυτή που ασχολείστε με την πρώτη μεγάλη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική η οποία μου είναι ιδιαίτερα προσφυλής όπως γνωρίζετε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε σε αρχή μίας εβδομάδας που ακολούθησε μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα με πολλή δουλειά. Με τον κύριο Τζοβάνι Τελαβία, με τον κύριο Καπούγια Σάντος και τον άλλο συναδελφό σας εργαστήκαμε πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε, εγώ ως πρώην Υπουργός γεωργία στη χώρα μου και τώρα υπάρχουν στην ενιαία ε, εσωτερική αγορά, πιστεύω ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να αφαισίσει την ποιότητα, στη διαφάνεια, στην ειχναλισμότητα και στην αηφορία. Κυρίε και κύριοι, αυτό το πρότυπο, το ευρωπαϊκό, για μένα θα πρέπει να ενισχυθεί σε σχέση με την αγορά. Με απέτηση ή αντικειμενικό στόχο να υλοποιήσει αυτά τα οποία είπα τους όρους που χρησιμοποίησα προηγουμένως. Δεδομένου ότι στις αγορές πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα, καταχρήσεις και προκλήσεις. Το μόνο ε, και πρώτο εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την ΚΑΤ σε σχέση με την αγορά είναι να έχουμε ένα πιο ανθεκτικό αγροτικό τομέα έναντι στην ε, κρίσεις, έναντι στα προβλήματα, στα, διακυμάνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε διάφορα μέσα και εργασία ρύθμισης και διακανονισμών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σωστά. Αυτά τα οποία λέγω σε εσά. Τα λέγω και στον συνάδελφό μου Ντατσιάν Σόλος, τον επίτροπο που είναι υπεύθυνο για την Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το να ενισχύσουμε λοιπόν το γρηγορικό πρότυπο σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε και όλη την διατροφική ε, αλυσίδα σε όλες τις συσφάσεις και όλες τις σχέσεις με όλους τους άλλους τομείς και προσπαθώντας να ρυθμίσουμε τις ε, τάσεις τις κερδοσκοπικές οι οποίες παρουσιάζονται εδώ και πολλά χρόνια και κάνουν τις τιμές ε, των βασικών αγαθών να εκτοξεύονται στα ύψη. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο με τα οποία ασχολούμαι ιδιαίτερα και τα οποία εγώ θα σας μιλήσω σήμερα. Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, βασικά αγαθά και την διατροφική αλυσίδα. Όπως ξέρετε, στην αλυσίδα ε, προμήθεια, την διατροφική ή όχι, στις 31 Ιανουαρίου εγκρίναμε μία πράσινη βίβλο, μετά από την οποία αρχισαμε μία εκτεταμένη συζήτηση για θέμητες εμπορικές πρακτικές που υπάρχουν, είτε διότι δεν υπάρχουν γραπτές συμβάσεις, είτε διότι αναδρομικά στις συμβάσεις υπάρχουν αλλαγές, είτε για να σταματήσουν οι εμπορικές σχέσεις που βασίζονται σε που έχουν πολλές φορές ένα καταχρηστικό χαρακτήρα. Όλες αυτές οι αθέμητες πρακτικές, όπως ξέρετε, πλήττουν στο τέλος αυτούς οι οποίοι είναι λιγότερο προστατευμένοι, αυτούς οι οποίοι δεν αμείβονται καλά. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να μας οδηγήσει στο να έχουμε σε αυτές τις για αυτές τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές κάποιες προτάσεις. Ευχαριστώ που και συγχωρείτε με αυτό το θέμα και στον τομέα ε, της ε, ε, αλυσίδας προμηθειών και διανομής, καθώς και στις ε, ε, βιομηχανίες της μεταποίησης, θα πρέπει να δούμε σε όλα τα επίπεδα τι συμβαίνει. Ο κύριος Μπόρκ, ο οποίος καλένει και ο κύριος ε, Τσόλο συμμετέχουν στο φόρουμ το οποίο δημιουργήθηκε το 2010 και πρότεινε τον ορισμό του τι θα πρέπει να είναι οι δίκαιες σχέσεις και στα πλαίσια αυτής της ομάδας εργασίας μελετούμε αυτό το θέμα των των εμπορικών πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη ποια είναι τα πρότυπα των βέλτιστων καλών πρακτικών και με ποιο τρόπο μπορούμε να ρυθμίσουμε την κατάσταση. Επίσης, όπως ξέρετε, μέχρι σήμερα οι επαγγελματίες του αγροτικού κλάδου δεν θέλησαν να ε, συμμετάσχουν ακόμη σε αυτό το θέμα στα πλαίσια του φόρου εμείς ε, συμφωνήσαμε εν μέρη να αποθέσει να τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο μηχανισμός και ελπίζουμε ότι όλοι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε έγκαιρα για να καταλήξουμε θετικά αποτελέσματα. Ελπίζω ότι θα πρέπει σε, λογικά, σε λογικό χρονικό διάστημα να καταλήξουμε σε μία συμφωνία μεταξύ όλων. Και το λέγω διότι αυτό είναι κάτι προς συμφέρον όλων, είτε βρίσκονται στην διατροφική αλυσίδα είτε σε άλλους κλάδους. Το θέμα επίσης των διαφόρων ρυθμίσεων με τις τράπεζες ώστε να μπορέσουν κάποιες πρακτικές και κάποιες συνήθειες όσον αφορά ε, την διαφάνεια οι τράπεζες επίσης να συμφωνήσουν για να παρέχουν σωστές υπηρεσίες στους ε, πελάτες, στους καταναλωτές. Πρότεινα λοιπόν να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και εσείς επίσης και το Συμβούλιο να νομοθετήσει για τέτοιο είδους θέματα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε τελικά αυτή την ε, συμβατική πρακτική να τη θέσουμε σε εφαρμογή. Όλοι όμως γνωρίζουν ότι αν αυτή η σύμβαση που θέλουμε να κάνουμε και όχι η υποχρέωση δεν γίνει, ώστε να μπορούμε να εποπτεύουμε την όλη κατάσταση, θα περάσουμε ε, σε αποφάσεις που θα λάβουμε μετά δια της νομοθετικής οδού. Αυτά όσον αφορά τον μηχανισμό αυτό αυτορύθμιση, αν μπορώ να τον ονομάσω έτσι. Επίσης θα πρέπει να γίνει και η μελέτη αντικτύπου για να δούμε ποιες είναι θα οι επιπτώσεις. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος των θεμάτων που ασχολούμεθα θα περιμένω τις ερωτήσεις σας. Δεύτερο θέμα με τον οποίο ασχολούμαι είναι το θέμα της διαθέτησης και της ρύθμισης της αγοράς των πρώτων υλών, των βασικών προϊόντων. Εγώ, ως ξέρετε, επίσης ασχολούμαι με τα θέματα τα χρηματοπιστωτικά. Έχουμε εδώ και τρία χρόνια με αυτό το θέμα ασχολούμαι. Έχουμε περίπου 35 ε, νομοθετήματα. Όπως ξέρετε, είμαστε εδώ και τρία χρόνια σε κρίση και ασχολούμεθα με το θέμα αυτό και της νέας αγοράς των χρηματοπιστωτικών αλλαγών. Πρόκειται για μέσα τα οποία διαθέτουμε, τα οποία προτείνω για να μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα τις ε, διάφορες αυτές ε, διακυμάνσεις των ε, αγορών σε όλους τους τομείς, στον ενεργειακό και σε άλλους τομείς, στον εμπορικό, ώστε να μπορέσουμε να αμβλύνουμε, για να μην πω να ελέγξουμε τις κερδοσκοπικές τάσεις οι οποίες διαμορφώνονται. Η Ευρώπη προοδεύει, ενεργεί και αυτά γίνονται βάση πρόοδου και ενεργειών μας που γίνονται από εμάς και από σας στα πλαίσια της νομοθετικής σας εργασίας. Δεν θα επιμείνω για τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων ως των τιμών όσον αφορά τις πρώτες και τα βασικά προϊόντα. Δεν θα επιμείνω στο θέμα επίσης των χρηματοπιστωτικών διακυμάνσεων στις ε, αγορές των βασικών προϊόντων από το 2008 και μετά πρέπει να πω ότι το 2012 έχουμε μεγάλη αύξηση της ε, τιμής των βασικών προϊόντων και κερδοσκοπικές τάσεις παντού, σε όλες τις αγορές. Γιατί λοιπόν και αυτές τις αγορές θα πρέπει να τις ε, εξετάσουμε διαφορετικά. Δεδομένου ότι δεν είναι όπως οι υπόλοιπες αγορές. Δεδομένου ότι αφορούν βασικά προϊόντα, βασικά αγαθά, τα είδη διατροφής το επίπεδο ζωής και ευημερίας όλων των χωρών και με βαρύνοντα τρόπο κυρίως τις χώρες που είναι σε ανάπτυξη. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα αστάθειες και να μην υποστούν κυρώσεις ή πλέον αδύνατοι. Όπως είχα διαπιστώσει εδώ και τρία χρόνια, όταν ήμουν υπουργό Γεωργίας στη χώρα μου, πρέπει να ενεργήσουμε και αποφάσισα να ενεργήσω χρησιμοποιώντας τα διάφορα μέσα τα οποία διαθέτουμε, τα οποία θα σας αναφέρω σύντομα. Πρώτα απ' όλα, το ΕΜΙΡ, το κείμενο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ πρόσφατα οι τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες εγκρίνατε, που θα τεθεί σε εφαρμογή από φέτος. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ε, μέσον που αφορά τα παράγωγα προϊόντα. Και πρέπει να σας πω ότι οι παγκόσμιες συναλλαγές για τα παράγωγα προϊόντα ε, είναι μονίμως της τάξεως των 600 δις εκατομμυρίων ετησίως. Και εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και δεν ξέρει κανείς τι κάνει ποιο. Επίσης υπάρχουν τα παράγωγα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στην αγορά πρώτων υλών Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικός αυτός ο κανονισμός, ο ΕΜΙΡ, με μία κεντρική ε, βάση δεδομένων, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται στο trade repository όπως λέγεται όλα τα παράγωγα αγροτικά προϊόντα ώστε να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια. Και σε αυτό τον κανονισμό των ΕΜΗΡ υπάρχει και η υποχρέωση ε, τυποποίησης ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα τυποποιημένα παράγωγα προϊόντα και κάποιες εγγύσεις για τα μη τυποποιημένα. Προσπαθούμε λοιπόν με το ΕΜΙΡ να βελτιώσουμε την κατάσταση και για να είμαι δίκαιο θα πρέπει να πω ότι δεδομένου ότι πρόκειται για απόφαση η οποία ελήφθη σε επίπεδο του G20 για τα αγροτικά προϊόντα. Όπως και είπα και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε εκ παραλλήλου. Δεύτερο μέσον, το MIFID, το οποίο είναι στο στάδιο της συζήτησης εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών. Πρόκειται λοιπόν για το ΜΥΦ, αυτή τη νέα οδηγία, ώστε ό,τι δεν είχε ακόμη ε, ρυθμιστεί εξαιτία αδυναμιών ή άλλων προβλημάτων να μπορέσει να ρυθμιστεί στις δημόσιες αγορές, ώστε να μπορέσουμε όλους όσους ε, ε, καλύπτονται στις δημόσια αγορές για αυτά τα παράγωγα προϊόντα να μπορούμε να τους έχουμε μέσα σε ένα κεντρικό πλαίσιο. Ελπίζουμε ότι αυτή η οδηγία θα μπορέσει να εγκριθεί χάρη και στις δικές σας εργασίες στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Τρεις δος άξονας να ενισχύσουμε του δεσμούς μεταξύ της εποπτείας των αγορών όταν είναι χρηματοπιστωτικές ή των αγορών ε, των άλλων ώστε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους των ε, φυσικών ας πούμε αγορών και των χρηματοπιστωτικών. Και εδώ χρησιμοποιούμε την οδηγία που αφορά τις ε, καταχρήσεις στην αγορά, που αφορά τις αγροτικές αγορές, την αγορά του φυσικού αερίου, ώστε να υπάρχει για όλους σωστή ενημέρωση. Τέταρτο μέσο, να μπορέσουμε τα μέσα εποπτείας να τα ενισχύσουμε. Και εδώ υπάρχει η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας ΜΥΦ ώστε να υπάρξει πρόεδρος ενισχύοντας τις εξουσίες των εποπτικών οργάνων υπό την εποπτεία της ΕΣΜΑ. Προτείναμε λοιπόν οι διάφορες ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο θέμα των παραγόγων προϊόντων, των αγροτικών προϊόντων και όταν χρειάζεται, και αυτό είναι σημαντική πρόοδος, την οποία πρότεινα και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ε, γνωρίζουμε πότε φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις ώστε να εμποδίσουμε κάποιες μονοπολιστικές ε, καταστάσεις σε κάποιες αγορές και κυρίως τις πιο ευαίσθητες. Αυτό λοιπόν είναι το τέταρτο μέσο μέσω αυτής της οδηγίας MIF ή κάποιες ε, ακραίες θέσεις ε, στις οποίες δεν θέλουμε να φτάνουμε όπως υπάρχει και σε άλλες υπήρους. Το επόμενο θέμα είναι η καταχρήση στην αγορά. Όπως σας είπα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στη διαπραγμάτευση και προτείνουμε να μπορέσουμε να δώσουμε τον ορισμό του. Τι σημαίνει για τα παράγωγα προϊόντα που αφορούν τις πρώτες ύλες κατάχρηση στην αγορά, ώστε διάφορες καταχρηστικές πρακτικές και συμπεριφορές να μην συμβούν και αυτό θα μας βοηθήσει να το κατορθώσουμε ύπαρξη της σωστής κοινοτικής νομοθεσίας. Ε, όλα αυτά τα θέματα ήταν θέματα τα οποία φάνηκαν τώρα με την οικονομική κρίση ε, και πρέπει να πω ότι κυρίως αναφέρομαι στην ε, χειραγώγηση κάποιων δικτών. Αυτόν τον κίνδυνο χειραγώγησης που αφορά την, στον τραπεζικό τομέα κυρίως τους δείκτες, κανένας δεν το είχε φανταστεί, υποψιαστεί. Κανένας δεν μας είχε προειδοποιήσει το ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και αυτό το συνειδητοποίησαμε, το είδαμε, με αυτά τα οποία έγιναν με τον δείκτη Labor, Libor, και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι Βλέπετε εδώ ποια είναι τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε και το χρονοδιάγραμμα και όταν ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας πρέπει να πω ότι κανένας τομέας και καμία αγορά δεν θα μπορέσει να εξαιρεθεί από τον ε, κανονισμούς στους οποίους θα πρέπει να τηρούν και να σέβονται. Ό,τι κάνουν θα πρέπει να γίνονται με διαφάνεια πολύ περισσότερη από ό,τι στο παρελθόν. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ε, χρηματοπιστωτικής ε, ρύθμισης και των ε, κανονισμών που αφορά κυρίως τα βασικά προϊόντα και κυρίως τις πρώτες ύλε που αφορούν την γεωργία και σας ευχαριστώ που με επιτρέψατε να λάβω το λόγο να σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ Μισελ. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητες τις οποίες έχεις και επίσης εμπιστευόμαστε την πολύ σημαντική γνώση που έχεις του γεωργικού τομέα. Είμαστε λοιπόν πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει σωστέ πρωτοβουλίε όσον αφορά για παράδειγμα το ζήτημα τη διακύμανση των τιμών, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Ξέρουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τη διακύμανση των τιμών έχει να κάνει με κερδοσκοπικέ τάσει στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Πρωτού δώσω το λόγο στους συναδέλφους και φαντάζομαι ότι ερμηνεύω πολύ καλά την θέληση όλων των συναδέλφων εδώ πέρα, θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμού μας, τη σκέψη μας όλων στον κύριο Παπαστάμκο. Η κατάστασή του είναι πολύ δύσκολη, αλλά ελπίζουμε ότι θα καταφέρει να επιστρέψει και να είναι σύντομα μαζί μας εδώ πέρα στην Επιτροπή Γεωργίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο Επίτροπος Μπαρνία πρέπει να φύγει στις 4. Συνεπώς, καθότι πρέπει να του δώσουμε 10 λεπτά για να απαντήσει, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι σύντομε οι παρεμβάσει σα, μέγιστο 2 λεπτά. Ξεκινάμε με την Πατρά Οντεβές και στη συνέχεια με τον ε, κύριο Νταντάν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί αναφερθήκατε σε δύο ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Επιτροπή Γεωργίας. Δεν έχουμε λοιπόν πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ πολύ γρήγορα στο πρώτο σημείο, τροφική αλυσίδα. Είπατε και έχετε απόλυτο δίκιο ότι η κοινή γεωργική πολιτική, προκειμένου να ενδυναμωθεί, πρέπει να ενδυναμώσει και όλη τη διατροφική αλυσίδα και αυτό αληθεύει. Γιατί οποιαδήποτε μεταρρύθμιση και να επιφέρουμε στην κοινή γεωργική πολιτική, αν δεν καταφέρουμε να έχουμε μία σωστή διανομή των εσόδων σε όλη τη διατροφική αλυσίδα, τότε στην πράξη η γεωργία σίγουρα θα ζημιωθεί και θα υποφέρει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Φεβρουάριο 2012 ένα ψήφισμα στο οποίο λέει ότι πρέπει κατεπηγόντως να εγκριθούν βέλτιστες πρακτικές ως προς την τροφική αλυσίδα και λέει επίση ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλυφθούν και νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Εμεί ακόμα περιμένουμε αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περιμέναμε ω τον Ιούλιο, γιατί ε, τον Ιούλιο το φόρουμ υψηλού επίπεδου λογικά θα πρέπει να καταλήξει κάποια συμπεράσματα. Στη συνέχεια περιμέναμε μέχρι τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και εν τέλει η Κοπάκα Κοζακά αποχώρησε από τη συμφωνία αυτή και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνία στο γεωργικό τομέα αν δεν έχουμε μέσα τους γεωργούς και συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πράσινη δίπλα. Εμεί περιμέναμε μια ανακοίνωση. Ειλικρινά σας λέω κύριε Πίτροπε ότι έχω απογοητευτεί από αυτή την κατάσταση. Μας μιλήσατε σήμερα για τον έφθετο αυτό χρόνο, τον λογικό χρόνο που απαιτείται προκειμένου να καταφέρουμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για συμβάσεις, αλλά εμείς μιλάμε εδώ πέρα και τέσσερα χρόνια για το ζήτημα αυτό και περιμένουμε τέσσερα ολόκληρα, ολόκληρα χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή να αρχίσουμε να μιλάμε επισήμω για μια ελάχιστη αν μη τι άλλο νομοθεσία, και να καταφέρουμε να καταλήξουμε και σε μια σύμβαση βελτίστων πρακτικών. Νομίζω ότι χρειάζονται και τα δύο, και η σύμβαση και η νομοθεσία. Το να μιλάμε αυτή τη στιγμή και να επενδύουμε μόνο σε σύμβαση βελτίστων πρακτικών θεωρώ ότι δεν μας ωφελεί και είναι και ιδιαίτερα χρονοβόρεια όλη διαδικασία. Ήδη έχουμε περιμένει πάρα πολύ. Ο Μισελ Νταντέν έχει τώρα το λόγο και στη συνέχεια η Ελίζα Γέγγελ. Κύριε Επίτροπε, πήρατε το λόγο λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την ψηφοφορία που έλαβε χώρα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα τέσσερα νομοθετήματα για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πραγματικά συμφωνούμε με τα όσα είπατε και εμείς ουσιαστικά ασχολούμαστε με τα ίδια ζητήματα. Είπατε ότι το να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τα παλαιότερα μέσα της κοινή γεωργικής πολιτικής για μια μελλοντική γεωργική πολιτική είναι κάτι το αδύνατο. Θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε νέα μέσα προσαρμοσμένα στη νέα κατάσταση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αναφερθήκατε επίση στο τι κάνουν τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρυθμίσουν τι αγορέ ε, πιστοτικών προϊόντων σε βασικά γεωργικά προϊόντα, τι γίνεται όμως για το ίδιο ζήτημα σε άλλες γωνιές του κόσμου. Γιατί αυτό που έχουμε συνειδητοποιήσει εμείς είναι ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια να ανταποκρίνεται στις απαιτήσει του G20, συνεδρίαση μάλιστα που έγινε κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας, οι ρυθμίσεις όμως αυτές στον τομέα των προϊόντων, των χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε βασικά γεωρικά προϊόντα δεν πρόκειται να αποδώσουν αν δεν ακολουθήσουν τις ίδιες απαιτήσεις και τις ίδιες ρυθμίσεις και οι υπόλοιπε χώρες του κόσμου, οι τρίτες χώρες. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίσουμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστούμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Ελίζαμπεθ Γέγκελ και ο Μάρκ Ταραμπέλα στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε στην συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής Γεωργίας. Μετά την ψηφοφορία που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, κάνατε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τη γεωργική πολιτική, αναφερθήκατε στη βιωσιμότητα, τη διαφάνεια, στην ιχνηλασιμότητα. Και θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω το εξής ερώτημα, εφόσον είστε Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς. Η γεωργία αποτελεί τμήμα της εσωτερικής αγοράς. Επομένως, ε, ποιο είναι το περιθώριο βελτίωσης που έχουμε όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα και τη διαφάνεια. Αν δούμε για παράδειγμα το σκάνδαλο με το κρέας ε, αλόγου, το οποίο έπληξε πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε και άλλα παραδείγματα, όπως για παράδειγμα τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει με τα αντιβιωτικά σε κάποιες περιπτώσεις τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στον τομέα της χνηλασιμότητας, πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα υψηλό επίπεδο χνηλασιμότητας για όλη τη διατροφική αλυσίδα με διαφανή τρόπο. Χάρηκα πάρα πολύ για τα θετικά δυναμικά σχόλια τα οποία κάνατε και για τα σχόλια τα οποία είπατε για τις ομάδες παραγωγών, λέγοντας ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένες διατάξεις. το σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, όπω είπατε και εσεί ότι δεν χρειαζόμαστε μια πλήρη απελευθέρωση του τομέα. Χρειαζόμαστε μια ρυθμισμένη, πλαισιωμένη αγορά στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς, η οποία θα διέπεται από συγκεκριμένου κανόνε. Αν μπορείτε να απαντήσετε στα ζητήματα αυτά, παρακαλώ. πρόεδρο. ευχαριστούμε πολύ. Μάρκ Ταραμπέλα είναι ο επόμενο ομιλητή. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα τη κερδοσκοπία. Διάβασα την το βιβλίο το οποίο γράψε όταν ήσασταν υπουργό Γεωργίας με τίτλο Ποιο θα θρέψει τον αυριανό κόσμο» θεωρώ ότι είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης αυτό το βιβλίο. Ειλικρινά σα το λέω. Και βλέπουμε ότι σήμερα πραγματικά πρέπει να θέσουμε το ζήτημα αυτό. Τα τροφικά γεωργικά προϊόντα είναι προϊόντα αλλά Ξέρω ότι ε, πολλές φορές ε, αποτελούν αντικείμενο διμερών συμφωνιών ή συμφωνιών στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι, για παράδειγμα, το 2010 μετά από φωτιές στην Ρωσία, πυρκαγιές στη Ρωσία, αυξήθηκε πάρα πολύ η τιμή του ΣΥΤΟΥ. Αντίστοιχες καταστάσεις είχαμε και για άλλα τρόφιμα, άλλα γεωργικά προϊόντα, τα οποία ήταν αντικείμενο κερδοσκοπία. Το 2010 επίσης στις παγκόσμιες αγορές 50 μπορούμε να πούμε φορές γίνανε ε, συναλλαγές όσον αφορά τον ΣΥΤΟ, την παγκόσμια παραγωγή ΣΥΤΟΥ. Νομίζω ότι θα πρέπει ουσιαστικά να μην είναι δυνατό να γίνονται οι συναλλαγές αυτές τη στιγμή που μιλάμε για βασικά γεωργικά προϊόντα και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μπορούμε να επιτρέπουμε να συναλλάσσονται στα χρηματιστήρια του κόσμου τόσος Τεράστιε ποσότητες γεωργικών προϊόντων. Καταλαβαίνετε, όταν αγοράζει κανεί 100.000 τόνους σίτου στι 9 ώρα το πρωί, μόνο και μόνο για να τι πουλήσει εκ νέου αυτέ, σε διαφορετική τιμή στι 4 ώρα το απόγευμα, υπάρχουν κάποιοι πληθυσμοί στον κόσμο που πληρώνουν ένα βαρύ τίμημα γι' αυτό. Επομένω, ποιε είναι οι δικέ σα παρατηρήσει και υπάρχουν ενδιασμοί ακόμα και στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σα ζητώ αυτή τη στιγμή να κατονομάσετε επιτρόπου οι οποίοι ενδεχομένω να μην θέλουν να ρυθμίσουν αυτή την αγορά. Θα ήθελα απλώ να γνωρίζω αν είναι ομοιογενή η στάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την κερδοσκοπία στα βασικά γεωργικά προϊόντα. Έχει μια κοινή στάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Πρόεδρο, ευχαριστούμε Μάρκα, Λεμπρού και Γκίρλινγκ είναι οι επόμενοι ομιλητέ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σας έχουμε δώσει στην Επιτροπή μας σήμερα. Πολύ περήφανοι, αλλά όχι ματαιόδοξοι. Επομένως, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε όλες αυτές τις θέσεις τις οποίες έχετε λάβει στο παρελθόν. Ήσασταν πάρα πολύ συγκεκριμένο ε, στα όσα είπατε. Θα ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη παρατήρηση και μια γενική παρατήρηση. Η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει να κάνει με τα μελλοντικά νομοθετήματα που θα μπορούσαμε να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον όπως είπατε και εσείς στο μέλλον ενδεχομένω η σύμβαση να μην έχει απόλυτα δεσμευτικό χαρακτήρα. Επίσης θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποια είναι η δική σας η άποψη για το ακόλουθο ζήτημα. Ποια είναι η γεωργία του αύριο. Ενδεχομένω να ακούγεται αφελέ το ερώτημα αυτό γιατί είναι πάρα πολύ γενικό αλλά θα ήθελα πραγματικά να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό. Ποια είναι η γεωργία του αύριο, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα μιλήσουμε επίσης και για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύετε ότι θα έχουμε τα απαραίτητα επαρκή μέσα, ότι θα έχουμε τις απαραίτητες δυνάμεις για να καταβάλουμε προσπάθειες κατά της απορριθμισμένης αυτής γεωργίας, που κάθε χώρα τελικά βάλει, κάθε μέρα, με συγχωρείτε, βάλει κατά της Ευρώπης θα είμαστε αρκετά δυνατοί ώστε να μην γίνουμε υπεργολάβοι της Ινδίας, της Κίνας και της Βραζιλίας. Ευχαριστούμε Γκίρλινγκ και Όσλινγκ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είπατε ότι επρόκειτο να προχωρήσετε σε μια διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την αγορά παραγόγων σε βασικά γεωργικά προϊόντα και θεωρώ ότι αυτό είναι θεμελιώδε. Μετά τα όσα είπε ο κύριο Νταντάν, θα ήθελα να θέσω το ακόλουθο ερώτημα. Θεωρείτε θεμελιώδε να έχουμε μια παγκόσμια προσέγγιση στη ρύθμιση αυτών των αγορών και να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε και τα όσα λένε οι διεθνείς, ο Διεθνής Οργανισμός Επιτήρησης των Χρηματοπιστωτικών Αγορών. Αξίζει να καταλήξουμε ουσιαστικά σε μια κοινή εποπτεία των αγορών αυτών κάθε φορά που θα απαιτείται κάτι τέτοιο. Είτε θα πρέπει να έχουμε εκ των προτέρων μια πάρα πολύ αυστηρή θέση, με ένα μηχανισμό ο οποίος θα είναι αδιάλακτος και όχι ευέλικτος λοιπόν. Μάρτιν Όστιν και Αγνιό στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στο ζήτημα της κερδοσκοπίας όσον αφορά τα βασικά γεωργικά προϊόντα. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που δεν έχει συζητηθεί. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, κοιτάξει την αύξηση των τιμών στους τελευταίους χρόνους και υπάρχει μια δυνατότητα να απαγορευτούν τελείως οι ε, εικονικές αυτές συναλλαγές επί των γεωργικών προϊόντων. Αναφέρθηκε ότι από τον κύριο Ταραμπέλα, αν δεν κάνω λάθος, ότι γίνονται συναλλαγές 50 κομμασαπλάσεις από την αξία του καλαμποκιού, επί παραδείγματι. Υπάρχει λοιπόν κάποια δυνατότητα να επέμβουμε και να παρέμβουμε, να, να παρέμβουμε, να απαγορεύσουμε. Οι Goldman Sachs και η Deutsche Bank ε, έχουν δώσει ε, μια τεράστια αύξηση στον, ε, στην αξία των συναλλαγών ε, για διάφορες βασικές τροφές ε, μέσα σε μια περίοδο από το 2003 μέχρι τώρα που δείχνει πολλαπλασιασμό της αξίας των προϊόντων αυτών. Επομένως, υπάρχει κάποιος λόγος να ρυθμίζονται αυτές οι αγορές και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναμένει ενδεχομένως αντίδραση από κάποιους εταίρους ή μπορεί ενδεχομένως να περιμένει και συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό. Ευχαριστούμε. Άγνιου και ο κύριος Αντιπρόεδρος Σεκεργέσκη μετά από λίγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα θέλατε να μας ε, τοποθετηθείτε προς το θέμα του ε, αλογίσιου κρέατος. Ε, δεν το αναφέρατε καθόλου, παρότι μιλήσατε για εχνηλασιμότητα κτλ. Εμείς στη Βρετανία αισθανόμαστε μεγάλη απογοήτευση από, τις, από την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθμίσει τα θέματα του, της εχνηλασιμότητας των τροφίμων και πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε μόνοι μας να τα έχουμε καταφέρει πολύ καλύτερα. Αλλά και ο κύριος Ταραμπέλα αναφέρθηκε σε θέματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και που έχουν δοκιμαστεί και εγώ νομίζω ότι οι αγορές των ε, παραγόγων σε σχέση με τα γεωργικά προϊόντα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γιατί γίνεται λοιπόν αυτή η κερδοσκοπία, γιατί υπάρχει προσδοκία ότι θα υπάρξει έλλειψη στην αγορά. Μόνο λοιπόν το περιμένει κανείς ότι θα αυξηθούν οι τιμές αρχίζει να ε, φυτεύει περισσότερα, να καλλιεργεί περισσότερα. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολλά λάθη έχει ξεπεράσει τα εσκεμένα, αλλά υπάρχει εν τέλει και κάποιος τελικός χρήστης, τελικός κερδοσκόπος και όπως είδαμε και με την περίπτωση της πατάτας, όταν παρεμβαίνουμε σταματάνε τα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να παρέμβουμε και επίσης ε, βλέπω ότι οι λύσεις ενδέχεται να μοιάζουν με τις λύσεις που είδαμε πρόσφατα στην ε, Κύπρο. Δηλαδή η λύση για τη διάσωση του ευρώ ήταν η ε, καταλήστευση των τραπεζικών λογαριασμών των αποτομιευτών. Ευχαριστώ πολύ, Συγκιέρσκη και μετά Λάιον. Πρόεδρε, γίνεται λόγος για δραστηριότητες σε πολλούς τομείς και υπενθυμίζουμε τη συνεργασία με τον Επιτροπό Φίσλερ στην ανάπτυξη της Πέθρου και την γεωργική πολιτική. Η πολιτική της συνοχής φεύγει από την Ήπεθρο δεν υπάρχει επαρκής συνοχή. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της υπαίθρου των γεωργών, πράγμα το οποίο προϊονίζεται πολλά προβλήματα για το μέλλον. Και επίση σε σχέση με την παρουσία των γεωργικών προϊόντων στι διεθνεί αγορέ. Υπάρχει μια κοινοτικοποίηση στην ευρωπαϊκή κοινοτική αγορά, η οποία είναι σημαντική μένα, αλλά η παγκόσμια αγορά ε, ε, αντιμετωπίζει πάρα πολλά προσκόμματα. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου τι πρέπει να κάνει στον τομέα αυτών και τι πρέπει να επαφηθεί στην ελεύθερη λειτουργία των αγορών. Χωρί να παρεμβαίνουμε βέβαια στα πάντα. Και επίση ένα άλλο ζήτημα, η ποιότητα, οι προδιαγραφέ, διότι οι συναλλαγές, οι εμπορικές συναλλαγές και η μη εφαρμογή σε αυτέ τι εμπορικέ συναλλαγέ. των ε, διατάξεων, των ευρωπαϊκών διατάξεων, των διατάξεων που έχει ορίσει η ίδια η Ευρώπη για τις προδιαγραφές ποιότητας, επιτρέπουν σε όποιο κράτος παραβλέπει αυτούς ε, τους κανόνες, παραγνωρίζει τους κανόνες αυτούς, να καταστρέφει τις αγορές. Και από αυτό θα χάσουμε όλοι. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τον έλεγχο και να αντιμετωπίσουμε τις ε, καταστάσεις αυτές οι οποίες ε, οδηγούν σε σημαντική ζημιά για το ένα κράτος ή το άλλο σήμερα, αλλά κάποια στιγμή τους πάντες θα πλήξουν τα προβλήματα αυτά. Για να μην μιλήσω για το πλήγμα, το σημαντικό πλήγμα, το πλήγμα το οποίο εφίσταται η ίδια η ποιότητα των προϊόντων και η δυνατότητα διακίνηση προϊόντων καλής ποιότητας μεταξύ των κρατών. Χωρίς συνεργασία λοιπόν μεταξύ των κρατών μας, το θα Το υπόλοιπο θα είναι αρνητικό για τους πάντες. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάιον για να ολοκληρώσει. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία και την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία και να στήσω την, ε, τα σχόλιά σας. Καταρχάς ως προς την ε, βελτίωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα παράγωγα. Ξέρετε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόσφατα διορίστηκε η Κρίστιν Τάκερ ως διάμεσολαβητή διαμεσολαβητής τιμών για τα γεωργικά προϊόντα για να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στις τιμές. Έχει η κυρία Τάκερ τη δυνατότητα να παρέμβει εάν φανεί να υπάρχει κατά, κατάχρηση, ε, καταχρηστική τιμή δηλαδή σε κάποια προϊόντα. Ίσως λοιπόν το μοντέλο αυτό θα άξει τον κόπο να το εξετάσουμε και να το ε, διαδώσουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί πολύ συχνά ε, επικοινωνούν μαζί μου γεωργοί για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τους ενδιάμεσους, από τις ε, μεγάλες εταιρείες της ε, ε, κατεργασίας των προϊόντων τους. Επίσης, είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται οι αγορές για να αντιμετωπιστεί, για να προληφθεί καλύτερα, να γίνει το hedging δηλαδή, σε σχέση με, την, με μια μελλοντική πτυτικότητα τιμών. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να το προβλέψουμε και να το ρυθμίσουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε ανεξέλεγκτο. Το κύριο ζήτημα πάντως είναι εάν η κερδοσκοπία δημιουργεί ή απλώς ενισχύει το πρόβλημα της πτυτικότητας στις τιμές. Νομίζω ότι ισχύει το δεύτερο. Η πτυτικότητα που χαρακτήριζε το 2009 σχέση με τα γεωργικά προϊόντα είχε να κάνει περισσότερο από ό,τι είδε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βασική ιδέα ότι ήταν η αγορά ε, σε ε, έλλειψη, και σχετικά έλλειψη προϊόντων και άρα αντίστοιχα επηρεάστηκαν οι τιμές των γεωργικών προϊόντων. Επειδή είχε γίνει η επιλογή, ε, αντί να παράγονται τρόφιμα, η γεωργία να στραφεί προς τα βιοκαύσιμα. Άρα λοιπόν αυτή η πτυτικότητα ε, δημιουργείται ή επιδεινώνεται από αυτήν την ε, κατάσταση. Επίσης η ΕΣΜΑ θα πρέπει να ρυθμίζει, να επιβλέπει, να εποπτεύει στις αγορές. Το είπατε κι εσείς. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που να δείχνουν ότι μπορούν κάποιοι κερδοσκόποι να φέρνουν σε αδιέξοδο μια αγορά. Γιατί αν παραδείγματι θέλει κανείς να, να, να αγοράσει και να επηρεάσει με την απόσυρση από την αγορά ε, σιτηρά, θα έπρεπε να έχει τεράστια συλλό για να μπορέσει να αποθηκεύσει και τα σιτηρά που θα αγοράσει προκειμένου να επηρεάσει τιμές. Ευχαριστώ πολύ. Καπλώς Σάντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα και εγώ να σας χαιρετήσω. Έχουμε από την Γαλλική Προεδρία πολύ καλές αναμνήσεις και ελπίζω ότι ο κύριος Επίτροπος με τον ε, τρόπο που εργάστηκε μας κάνει όλους να ελπίζουμε ότι θα τον ακολουθήσουμε για να είμαστε σωστοί. Αυτά τα οποία μας είπατε μας φαίνεται πολύ συνεκτικά και λογικά. Ξέρω ότι τώρα ασχολείστε με την νέα εσωτερική αγορά, αλλά είσαστε πρώην Υπουργό Γεωργία. Διερωτώ όμω, εάν ε, ό,τι κάναμε το κάναμε σε συνεργασία με τους κύριους ε, ε, εμπορικούς συνεργάτες μας και εταίρους μας δεν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα παγκοσμίω, δεν θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Αναφέρομαι κυρίως στο θέμα του δίκτυ του Λίμπορ που είπατε. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε Λουίς, σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν σύντομοι στις παρεμβάσεις σας. Το λόγο έχει ο Μισελ Μπαρνιέ. Ε, για να απαντήσει. Να ακούσουμε και τον κύριο Ντόντε αν θέλετε. Να απαντήσει αυτό αντί για μένα αν προτιμάτε. Αλλά τέλο πάντων ο καθένα στη θέση του. Εφού ετάχθη. Και α μπερδεύουμε καμιά φορά τα ονόματα. Ή α συμφωνούμε σε ορισμένα θέματα. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ενώσω τη φωνή μου στι ε, ευχές για ταχύ αποκατάσταση ε, τον κύριο Γιώργο Παπαστάμκο, Έλληνα Ευρωβουλευτή. Όπως εκδηλώστηκε σε μέρους της Επιτροπής σας, έτσι και εγώ θα ήθελα ελπίζοντας ε, να ξεφύγει γρήγορα από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα. Εν συντομία θα απαντήσω. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις, για τα ενάψματα που μου δίνετε, για τις ερωτήσεις σας. Η κυρία Λεβέσκη, η κυρία Λεμπρά αναφέρθηκαν στην τροφική αλυσίδα. Πολλοί συνάδελφοί σας ανησυχούν. Όσο Ζεμποβέ έχει κάνει έκθεση για το θέμα αυτό. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, η κυρία, ο κύριος Γιούγκ έχουν ε, παρακολουθήσει εκ του σύνεγγες τα θέματα αυτά σε άλλες επιτροπές. Και πάλι θα μιλήσω περίφραστα Γνωρίζω ότι αθυμονείται. Πολλοί εξημών έχουν ήδη αποστείλει το στο γραφείο μου ζητώντα, να επιταχύνω την υποβολή νομοθετικών προτάσεων προκειμένου να πλαισιωθούν οι πρακτικές, να καταλήξουμε δηλαδή σε μια βελτίωση των πρακτικών των σχετικών με τροφική αλυσίδα και κυρίως με στόχο την προστασία του παραγωγού εγώ ιδιαίτερα με για το θέμα αυτό. Εργάζομαι όμως σε ένα συλλογικό όργανο, πέραν του γεωργικού παραγωγού ή του αμπελοϊνικού παραγωγού, του αμπελουργού. Έχουμε και άλλους φορείς, παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτή τη μακρά αλυσίδα της διατροφής. Τον κύριο Ντόντα, εξάλλου, έχουμε ήδη συζητήσει την σοβαρή αυτή ε, μετατροπή της αλυσίδας, ε, την αλλαγή της αξίας, την αύξηση της ε, αξίας, την προστιθέμενη αξία, που βέβαια σχετίζεται και με όλα τα τεχνικά ζητήματα και τις νέες απαιτήσει σε σχέση με την ποιότητα στο τρόφιμα, με θεμητά βέβαια αίτια και γνωστά πάντως αίτια, αυξάνει η τιμή μέσα σε αυτή την, ε, την ε, τροφική αλυσίδα και αντιλαμβάνομαι ότι όποιος βρίσκεται στην αρχή στο τέλος ε, της αλυσίδας αλλά κυρίως στην αρχή είναι, λιγότερο, είναι αυτός που εισπράττει λιγότερα, αμείβεται λιγότερο δηλαδή ή είναι λιγότερο προστατευμένος. Άρα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια για πραγματική πρόοδο στο θέμα αυτό και πριν από μερικές ημέρες στο Στρασβούργο και με τους εκπροσώπους της Eurocommerce, με τους οποίους έχουμε συνεργασία, έχω επισήμανα ότι δεν έχουμε απεριόριστη υπομονή. Δεν θα περιμένουμε επαόριστον. Κάνουμε τη δουλειά μας στο βαθμό που η αυτορύθμιση φέρνει αποτελέσματα κυρίως όσον την βελτίωση των συμβάσεων με τους προμηθευτές, τη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών κανόνων για βέλτιστη πρακτική ε, μεταξύ των παραγόντων της αγοράς ε, έχει καλός, αλλά και εμείς κάνουμε μελέτες ε, συνεπειών αξιολόγηση, το λεγόμενο αυτό twin track, όπως το ονομάζουμε, δηλαδή τον, την παράλληλη οδό και για να καθησυχάσω και την κυρία Λεμπρόν και την κυρία Λεμπρές, θα έλεγα ότι πολύ γρήγορα θα γίνει αυτή η μελέτη μέσα στο έτος, μέχρι το φθινόπωρο, εν πάση τους προσεχείς μήνες, θα αξιολογήσουμε τη λειτουργία του μηχανισμού, τις θετικές του πτυχές, εάν υπάρχουν, την χρησιμότητά του, εάν υπάρχει, γιατί δεν παίζουν όλοι σωστά με τους κανόνες και αν αυτό διαπιστωθεί, τότε θα εισαγάγουμε και τους κανόνες από πλευράς μας. Αυτή είναι η διπλή, παράλληλη δηλαδή πορεία την οποία έχουμε χαράξει. Είμαστε έτοιμοι να νομοθετήσουμε και πρέπει και εσείς να είστε από πλευρά σας εφόσον αποδειχθεί ότι έχει αυτή η ε, ενδοτική ε, λύση ε, αποτύχει. Γιατί δεν είμαστε αφελείς. Για την Κοτζέκα, με την οποία πάντοτε είχα σχέση και επικοινωνία, ελπίζω ότι θα μπορέσει να αναλάβει το ρόλο της και να μας βοηθήσει στην επαλήθευση του αν λειτουργεί ή όχι αυτός ο μηχανισμός. Και πάντως με τον κύριο Τσόλος πολύ ευχαρίστω θα, θα σας αναφέρουμε τα πορίσματα αυτής της μελέτης ε, αποτελεσματικότητας του μηχανισμού. Πάντως δεν θέλουμε να αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη του. Θέλουμε πραγματική πρόοδο στις σχέσεις με τους λοιπούς παράγοντες. Ο κύριος Νταντάν τώρα, ο κύριος Καπλασάντος, η κυρία Κιάνιν επεσήμαναν ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα ζήτημα πραγματικό, υπαρκτό, σε σχέση με το level playing field. Τι κάνουν λοιπόν οι άλλοι σε αγορές παγκόσμιες. Αυτό το level playing field όπως λέμε, δηλαδή το πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού, το μελετάω τακτικά και συνεχώς για να δω και τι κάνει η Ευρώπη αλλά και τι πράττουν οι υπόλοιποι, οι κύριοι εταίροι μα, οι Ηνωμένε Πολιτείε κυρίω, γιατί υπενθυμίζω ότι σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικέ αγορές και συναλλαγέ, το 80-80% των συναλλαγών, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, είναι διατλαντικού τύπου μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών. Δεν θα συνεχίσει στο δίνεκέ αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλε αγορέ. Δεν πρόκειται για την ε, Ασία, ειδικότερα για την Κίνα, το Χονγκ Κόνγκ, τη Σιγκαπούρη, ε, που αναδύονται και θα τραβήξουν ε, συναλλαγέ προ τα εκεί. Αλλά πάντω αυτή τη στιγμή έχουμε 80% στι διατλαντικέ συναλλαγέ. Κύριο Νταντά, κυρία Ντεγκαρίγα και κύριο Κάπουλα Σάντο, λοιπόν, νομίζω ότι αυτό εννοούσαν, αν καταλαβαίνω σωστά τι παρατηρήσει του. Έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μα εργαλεία, το EMIR, το MIFID, η, οδηγία σχετικά με την κατάχρηση των αγορών, ε, οι Αμερικανοί με, την, ε, με τη λεγόμενη dot Dodd-Front έχουν εισαγάγει παρόμοια μέτρα. Μερικές φορές μάλιστα ήταν και πιο προστατευτική από ότι εμεί σε σχέση με το ΕΜΗΡ με κάποιες ε, διατάξει περί διάθεσης στην αγορά των γεωργικών προϊόντων. Κάπου ήμασταν εμεί ε, πιο, ε, είχαμε εμεί πιο προωθημένε λύσει. Έχω ζητήσει πάντω από τι υπηρεσίε μου να κάνουν μια ειδική συγκριτική μελέτη και μάλιστα όχι μόνο σύγκριση μεταξύ του τι πράττουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, αλλά να βάλουν στον πίνακα και του Καναδού και του Βραζιλιάνου, του Ινδού, τους Κινέζους, τους μεγάλους δηλαδή παράγοντες και τους Ρώσους ακόμα, τους μεγάλους, ε, τις μεγάλες χώρες του G20, για να δούμε τι κάνουν. Θα σας διαθέσω, εφόσον το επιθυμείτε, τη μελέτη αυτή, τα πορίσματά της, μόλις τα έχουμε στη θέσή μας. Ε, πάλι στο μέτρο του δυνατού προχωρούμε. Πρόκειται για μια συγκριτική μελέτη μέσα στο πλαίσιο βέβαια των χρηματοπιστωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά πάλι στο πλαίσιο το περιορισμένο της ε, ρύθμιση των αγορών σε σχέση με την κερδοσκοπία που μπορεί να αφορά τα γεωργικά προϊόντα. Στο δε Μισελ θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερα επαγρυπνούμε σε σχέση με τις εργασίες της FAO, η οποία επίσης έχει ξεκινήσει από πλευράς της πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες, κυρίως όσον αφορά τη διαφάνεια. Τέσσερις τομές, τομείς στα σιτηρά, Ε, αραβόσιτο, σόγια, όριζα και στάρι έχουν ε, καλυφθεί από σχετικές μελέτε τη FAO, μελέτε που θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμε. Περιμένουμε να δούμε τα πορίσματά του. Και μια και συζητούμε αυτά τα θέματα τη παγκόσμια διακυβέρνηση ουσιαστικά, πάντα με προσοχή παρακολουθούμε τα, τις προτάσεις που ακούγονται σε επίπεδο FAO ή προς την FAO καλύτερα για μεταρρύθμιση για μια διαφορετική διαχείριση, διακυβέρνηση στον χώρο ιδιαίτερα της, ε, των τροφίμων και της γεωργίας. Τουλάχιστον αυτά τα είχα ήδη δει και από την προηγούμενη μου, τα προηγούμενα μου καθήκοντα. Επίσης ακούστηκε το θέμα της ίχνηλασιμότητας από κάποιους συναδέλφους. Ε, την λέξη αυτή την ε, χρησιμοποίησα και εγώ στην ομιλία μου νωρίτερα. Και θα αναφερθώ σε μια απάντηση σε μια αίθουσα, δεν θυμάμαι, μάλλον στο Στρασβούργο ήταν στην πρώτη μου ακρόαση υποψήφιο υποψήφιος ε, επίτροπος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες με την κυρία Λούλινγκ που δεν τη βλέπω σήμερα εδώ. Μου είχε ρωτήσει για το κρασί. Α, είστε εδώ, με συγχωρείτε. Με έχει στιγματίσει η κυρία Λούλινγκ. Με έχει σημαδέψει. Είχα κάνει λοιπόν αυτή τη σύγκριση, θα θυμάστε σας κυρία Λούλινγκ, για την ιχνηλασιμότητα μεταξύ των αμπελοϊνικών προϊόντων και των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ξεκινούσα ακόμα, δεν είχα καν να λάβει καθήκοντα ω επίτροπος επισήμω. Εγώ νομίζω όμως ότι υπάρχει δυνατότητα να ε, κάνουμε τον παραλληλισμό, γιατί πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συνεργασιμότητα και στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Σα είπα τι είδου μέτρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε για την συνεργασιμότητα. Πρέπει να ρίξουμε απλό το φω σε όλου αυτού που δεν είναι συνηθισμένοι να στέκονται στο φω, που δεν του αρέσει το φω στι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Ε, παραδείγματι, ο κανονισμό ΕΜΗΡ για τα παράγωγα προϊόντα θα αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση. Και σα υπενθυμίζω ότι και οι Αμερικανοί κάνουν κάτι αντίστοιχο εδώ τώρα ο γεωργός, ο παραγωγός, δεν έχει πρόβλημα με την ιχνηλασιμότητα, δεν ε, φοβάται την ιχνηλασιμότητα. Η κυρία Γέγκλο, ο κύριος Αγνιού, επίσης, εάν μιλάμε για την πρόσφατη κρίση, που σχετίζεται με απάτη, ξεκάθαρα, απάτη ως προς την φύση του προϊόντος που πωλήθηκε, αν ήταν δηλαδή βόηο κρέας ή ε, κρέας υποειδούς. Νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς άτεκτος έναντι όλων αυτών που αποτολμούν τέτοιες απάτες. Δεν διστάζω να πω ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι τέρματος της απέτηση για την ιχνηλασιμότητα όταν λέμε ότι πουλάμε βόηο κρέας στον καταναλωτή με τον ίδιο τρόπο και στο χρηματοπιστωτικό προϊόν πρέπει να υπάρχει μέχρι εσχάτων αυτή η ιχνηλασιμότητα. Και όπως είπα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να διστάζει από τους παραγωγούς να καταγράφεται το ίχνος του προϊόντος μέχρι και τελευταία, το τελευταίο στάδιο, το πακεταρισμένο δηλαδή ε, γεύμα. Και πρέπει να γνωρίζουμε ποιος αγοράζει τι και ποιος πουλάει τι, γιατί και αυτό συμβάλλει στην λασιμότητα. Κύριε Άγνιου, δεν θα τοποθετηθώ για την Κύπρο, που θίξατε εσείς νωρίτερα παρά μόνο για να πω ότι συνεχίζουμε τη συνεργασία με τις αρχές της χώρας εν ώψη της απόφασης που θα λάβει αύριο με την ψηφοφορία της η Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτή την άκρος έκτακτη και συνήθιστη απόφαση για την στήριξη των καταθέσεων και τη διαφοροποίηση που πρέπει να γίνει σχέση με τους μικροκαταθέτες. Αυτή είναι η δική μου θέση, αυτή είναι η θέση που με ως Ευρωπαίος Επίτροπος. Για τον κύριο Ταραμπέλα, τον κύριο Χόισλινγκ. Αναφερθήκατε και ιδίω ε, στην κερδοσκοπία. Κύριε Ταραμπέλα, ερώτηση, αν πρέπει να απαγορευτεί. Κοιτάξτε, μπορεί να έχει κάποια χρησιμότητα για την κυκλοφορία της, ε, του ρευστού αυτές τις συναλλαγές. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν ζητήσαμε. Άλλωστε και το Κοινοβούλιο σε κάποιους τομείς μας υποστήριξε. Δεν ζητήσαμε απαγόρευση, πλήρη απαγόρευση. Όμως, κύριε Ταραμπέλα, πιστεύω, όπως και εσείς, ότι χρειάζεται πολύ αυστηρή πλαισίωση ως προς, τις, ε, ως προς τα όρια των ε, θέσεων και ίσως θα έπρεπε να είναι και εξάντε, εκ των προτέρων δηλαδή τα όρια, όχι μόνο εκ post, εκ, post, εκ των υστέρων. Οι εξουσίες της ΕΣΜΑ θα είναι ε, να αποφασίζει όταν υπάρξει κίνδυνος έκρηξης, πτυτικότητας, που διαπιστώθηκε και στο παρελθόν με σοβαρότατες συνέπειες ως προς τη σταθερότητα, αλλά ακόμη και την ασφάλεια της ε, προμήθησης τρόφιμα, να επιβάλλει ξεκάθαρα όρια σε αυτές τις θέσεις για τον κύριο Χόισλινγκ, για να μπορέσουμε να ποσοστοποιήσουμε όπως το ζητάτε και όπως και εγώ θα πω το επιθυμώ, πρέπει να γνωρίζουμε επακριβώ, πρέπει να έχουμε υπόψη και γι' αυτό η υποχρέωση της διαφάνειας που έχουμε συμπεριλάβει στο κείμενο, για τη μύφιντε παραδείγματι, αλλά και για την εμίρ, για τα παράγωγα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με προϋποθέσεις για την ποσοτική αξιολόγηση αυτών των φαινομένων. Πρέπει να ξέρουμε ποιος κάνει τι, γιατί την ποσοστοποίηση δεν μπορούμε να την κάνουμε ε, εάν δεν γνωρίζουμε ποιος έχει αγοράσει τι ή ποιος έχει προβεί σε ποια συναλλαγή. Πάντως η κατεύθυνση που ακολουθούμε είναι η ίδια. Τον κύριο Σκέσκι δεν σας λησμόνισα και τη δυνατότητα δηλαδή ε, για την συνέχιση της πολιτικής της συνοχής δεδομένων και των προηγουμένων καθηκόντων του Επιτρόπου για τα περιφερειακά θέματα. Η συνοχή έχει πολύ μεγάλη σημασία για την γεωργική πολιτική, ιδιαίτερα στο δεύτερο πυλώνα και γι' αυτό και υποστηρίζω τον κύριο Χάν, τον συνάδελφο Γιωάννης Χάν, ε, στις προσπάθειές του αυτές, με την ελπίδα ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο βέλτιστο δυνατό προπολογισμό όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις που ξεκινούν μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ώστε να ε, στηριχθούν αυτές οι δύο πολιτικές, οι οποίες δεν είναι επεπαλαιωμένες, δεν είναι απαρχαιωμένες πολιτικές, δεν ανήκουν στο παρελθόν, είναι σύγχρονες πολιτικές και απαραίτητες, τόσο η γεωργική όσο και η πολιτική της συνοχής. Για τον κύριο Σικέσκι θα ήθελα να επισημάνω ότι βεβαίω και θέλω πολυμερει συμφωνίες σε σχέση στον τομέα του εμπορίου στα γεωργικά προϊόντα. Πάντα θεωρώ ότι είναι καλύτερες. Ξέρω γιατί και δεν ξεχνάω ποτέ γιατί απέτυχαν οι τη ΔΟΧΑ λόγω της ε, απουσία συνένεση, ή μάλλον συμφωνία με του Αμερικανού, με την Αμερικανική πλευρά. Πρέπει να συνεχίσουμε, αλλά εν αναμονή των ε, αποτελεσμάτων σε πολυμερέ επίπεδο, στον ΠΟΕ συνεχίζουμε τι διμερεί επαφές με τους Καναδούς, πάνε αρκετά καλά, με του Αμερικανούς προσταθούμε χωρί βέβαια να είμαστε αφελεί ε, και να ε, περιμένουμε ιδεώδεις λύσεις, είμαστε ενεργοί στις διαπραγματεύσεις, περιμένουμε ίσως με την ε, με κάποιες εξελίξεις από πλευράς αμερικανικής να συμπεριληφθούν και τα γεωρικά προϊόντα. Κύριε Λάιον. Ε, στις ε, παρατηρήσεις σας σε σχέση με αυτό το όργανο εποπτείας ή ελέγχου των τιμών σε περίπτωση καταχρήσεων. Ε, πρέπει να επισημάνω ότι είναι βρετανικό το παράδειγμα που μας δώσατε, ειδικά βρετανικό, αλλά αντίστοιχο ρόλο μπορεί να αναλάβει η ΕΣΜΑ και αντίστοιχα να παρεύουν και οι εθνικές ε, εποπτικές αρχές. Αλλά θα το κοιτάξουμε πιο προσεκτικά αυτό που προτείνεται. Θα μελετήσουμε δηλαδή τι ακριβώς σύστημα ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αξιοποιήσουμε οι δυνατόν τα διδάγματα αυτού για τον κύριο Λάιον ή τον κύριο Κάπλο Σάντος που ίσως είχε επισημάνει το θέμα της βράχυπρόθεσμης πτυτικότητας των τιμών και ζητήματα που σχετίζονται είτε με τις ε, κλιματικές αλλαγές είτε με τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Ε, είναι ασφαλώς συνέπεια άμεση και ξεκάθαρη που όμως ε, οξύνεται σε φαινόμενο από τη λειτουργία των αγορών. Στη δε υπόθεση που αναφέρατε νωρίτερα, και η κυρία Γέκλη και ο κύριο Άγνιου για το κρέα αλόγου αντί για το βόλιο κρέα στην τροφική αλυσίδα. Ε, πρέπει να μελετήσουμε ακόμη περισσότερο την αλυσίδα, γιατί υπάρχει μια διαδικασία ολόκληρη τη οποία δεν έχουμε αντιληφθεί κάθε λεπτομέρεια. Υπάρχει κάποιο, υπάρχουν κάποιοι παράγοντε, κάποια στοιχεία αυτή τη αλυσίδα που είτε οδηγούν είτε ενισχύουν τον κίνδυνο τη απάτη ή τα αποτελέσματα τη απάτη καλύτερα. Και αυτό ακριβώ αυτή η μετατροπή σε χρηματοπιστωτικέ των αγορών αυτών των πρώτων υλών ε, είναι που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγάλη, με μεγάλη προσοχή. Εμεί είμαστε αποφασισμένοι, ε, στηριζόμαστε και στη δική σα αποφασιστικότητα για την έγκριση και των κειμένων που ήδη πρόσφατα εγκριθήκαν όπω το ΕΜΗΡΙ που θα πρέπει ε, σχετικά σύντομα να εγκριθούν όπω το ΜΥΦΙΔ ή η η οδηγία για τι αγορέ. Εν πάση περιπτώσει θέλουμε τα μέτρα αυτά που θα μα επιτρέψουν και την ανεχνευσιμότητα και την διαφάνεια στις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικέ αγορές για πρώτες ύλες γεωργικού, γεωργικής προέλευσης να εξασφαλίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σταματώ σε αυτά και δεσμεύομαι κύριε Πρόεδρε σε μερικούς μήνες να επανέλθω και να σας ενημερώσω όταν θα έχουν υιοθετηθεί και αρχίσει να εφαρμόζονται τα σχετικά νομοθετήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε, αγαπητέ φίλε Μισελ Μπαρνιέ. Νομίζω πραγματικά ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Επίτροπο, ο οποίος ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Και βέβαια προφανώ και εμά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να παρακολουθήσουμε τις εργασίες Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στο μέλλον για τα σημαντικότατα αυτά ζητήματα. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ πολύ. Περάσαμε λίγο το χρόνο το οποίο προβλεπόταν. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστούμε Μισελ Μπαρνιέ. Ένα λεπτό διάλειμμα. Allora Ας συνεχίσουμε, παρακαλώ, τις εργασίες μας. Colleghi, Ας συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα μετά το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, Στη συνέχεια έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με μέλη του ε, τμήματος 1 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 5 η ώρα. Γρήγορα λοιπόν να σκαλύψουμε το σημείο 5 και στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι να φτάσουν τα μέλη από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, Αγροτικέ και λευτικέ στατιστικέ, αγαπητοί συνάδελφοι, α περάσουμε τώρα στην εξέταση του σχεδίου έκθεση επί τη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόταση κανονισμού το οποίο τροποποιεί ορισμένε νομοθετε... ορισμένες νομοθετικές πράξεις στον τομέα των αγροτικών και λευτικών στατιστικών. Εγώ είμαι συγητή για την έκθεση αυτή. όπω ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε, σύμφωνα με τον κανονισμό 182 του 2011, να επανεξετάσει με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στη συνθήκη όλες τις πράξεις που περιέχουν αναφορές στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Ο γενικός στόχος είναι μέχρι το τέλος της 7ης θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο 2014, να εξαλειφθούν οι διατάξεις και να υποκατασταθούν από κατεξοδότηση πράξη. Στόχο τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να τροποποιηθούν 9 νομοθετικέ πράξει στον τομέα των γεωργικών και λευτικών στατιστικών, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Ένα δεύτερο στόχο τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο εξορθολογισμό του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αντικατασταθεί η αναφορά στη μόνιμη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών με μία αναφορά σε μία άλλη Επιτροπή, δηλαδή την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, που όπως θυμάστε θεσπίστηκε με τον καονισμό 223 του 2009 και θεωρείται ως το ανώτερο στρατηγικό όργανο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Η Επιτροπή αυτή επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών σε, ορισμένου στατιστικού τομεί. στατιστικούς τομείς. Ως θεωρώ ότι ε, το κείμενο αυτό δεν παρουσιάζει προβλήματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο βασικός στόχος είναι να αντικατασταθεί η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο με κατεξοδότηση πράξη και στα εννιά νομοθετήματα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιπτώσεις της παλαιάς λεγόμενης επιτροπολογίας, που παραμένουν ως εφαρμοστικά μέτρα, θεωρώ ότι δεν αποτελούν πρόβλημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι πρόκειται για έντυπα διαβίβασης τελικά ή πολύ συχνά για απλές παρεκκλήσεις για ορισμένα κράτη-μέλη. Πρόκειται ουσιαστικά για διατάξεις οι οποίες ε, ουσιαστικά καλύπτονται από εκτελεστικές πράξεις. Καταλήγοντας, κατέθεσα εννέα ταυτόσιμες τροπολογίες, μία για κάθε νομοθετική πράξη, προκειμένου να επαναφέρω τη διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στα θεσμικά όργανα όσον αφορά τις κατεξοδότηση, τις κατεξοδότηση πράξης. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι η περίοδος εξοδότησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι αόριστη, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται σε μία πενταετή περίοδο. Προτού δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Υπηρεσιών. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο συνάδελφο που θέλει να πάρει το λόγο πριν τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν όχι, δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Μαρσέλ Ερμέν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που δίνετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για την πρόταση αυτή η οποία έχει ως στόχο όπως το τονίσατε κι εσείς να καταφέρουμε για τα εννέα αυτά νομοθετήματα, για τις εννέα αυτές νομοθετικές πράξεις, για τις γεωργικές και ελευθερικές στατιστικές, να ευθυγραμμιστούν τελικά με τις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Στόχος μας λοιπόν είναι, μέχρι του χρόνου ή δυνατόν, να αφαιρέσουμε όλες αυτές τις διατάξεις που αναφέρονται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, από τα 9 αυτά νομοθετήματα, από τις εννέα αυτές νομοθετικές πράξεις. Αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Ο δεύτερος στόχος, όπως το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, είναι να αντικαταστήσουμε την επιτροπή αυτή η οποία ήταν αρμόδια για τη διαδικασία επιτροπολογίας στις εννέα αυτές νομοθετικές πράξεις που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι ακόμα η μόνιμη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον τον κανονισμό 223 του 2009, ο οποίος αναφέρεται πλέον σε ένα ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα. Θέλουμε να καταφέρουμε να ευθυγραμμίσουμε τι στατιστικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θέλουμε να ενισχύσουμε το πλαίσιο εκείνο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει καλύτερες εταιρικές σχέσεις ανάμεσα στις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή τη Eurostat. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε καλύτερα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η μόνιμη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών θα πρέπει να αντικατασταθεί από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, όπως ακριβώς κάναμε δηλαδή και με άλλους τομείς παροχή στατιστικών υπηρεσιών. Θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να εξορθολογήσουμε καλύτερα τα όσα προκλεπόντουσαν στην παλαιότερη διαδικασία επιτροπολογία. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το αργότερο μέχρι του χρόνου, μέσω του 2014, θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και όλος ιδιαίτερος θέλω να σε ευχαριστήσω εσάς κύριε Πρόεδρε γιατί αποδεχτήκατε να είστε ο εισηγητής για την έκθεση αυτή. Προέδρο, ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχουν άλλε παρατηρήσει, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 21 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι. Αν δεν υπάρχει κανεί άλλο που θέλει να πάρει το λόγο, α κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τι 5. Στι 5 θα φτάσουν στην Επιτροπή μα, οι προσκεκλημένοι μα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να μα ενημερώσουν για την κοινή γεωργική πολιτική. Διάλειμμα λοιπόν μέχρι τι 5. Bene, colleghi, possiamo iniziare. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πρόεδρο και τα μέλη του πρώτου τμήματος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που ασχολούνται με ζητήματα διατήρησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Ιωάννη Σαρμά, την κυρία Ράζα Μπούτγκερ Μπάιτ, τον κύριο Μισελ Χαϊτάν και τον Αγγουστίν Κούμπικ. Καταρχά, θα έχουμε μια σύντομη εισαγωγική δήλωση για τι εργασίε του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και ιδίω την εργασία που κάνει το πρώτο τμήμα και στη συνέχεια θα ακούσουμε μια παρουσίαση τη γνώμη του Ελεκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τι προτάσει μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική με κάποια σχόλια όσον αφορά τι τροπολογίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο τέλο, θα ακούσουμε τι έχει δηλώσει το Ελεκτικό Συνέδριο στι εκθέσει του όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, την γεωργοπεριβαλλοντική πολιτική, την αποσύνδεση και την ανάπτυξη τη υπαίδρου. Θα έχουμε στη συνέχεια μια ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους του Ελεκτικού Συνεδρίου και δίνω ευθύς αμέσως το λόγο στον πρόεδρο του πρώτου τμήματος, ευχαριστώντας τον ίδιο, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου που είναι σήμερα μαζί μας και θα καταφέρουμε από κοινού κατά αυτόν τον τρόπο να συζητήσουμε τις δικές σου παρατηρήσεις. Κύριε Σαρμά, έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε να μας υποδεχθείτε σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σημερινή συνάντηση στις τρεις είναι πολύ απλή ιδέα. Το τμήμα μας, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, ε, ασχολείται με θέματα και προβλήματα στην γεωργική ανάπτυξη και την ανάπτυξη πέθρου, που ενδιαφέρουν βέβαια και την δική σας Επιτροπή. Θα ήταν χρήσιμο για τις δύο πλευρές πιστεύω να ανταλλάξουμε απόψεις ως προς τις κύριες ε, ιδέες μας ή τα κύρια, τις κύριες διαπιστώσεις ως προς ε, τη γεωργία και την ε, ανάπτυξη πέθρου. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι μοιρασμένο σε πέντε τμήματα. Αυτό που ασχολείται με την γεωργία και την ανάπτυξη της πέθρου είναι το πρώτο απαρτίζεται από έξι μέλη. Σήμερα ήρθαμε τέσσερις. Ο ένας είναι ασθενής και ο άλλος είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση και δεν μπόρεσε να έρθει. Ο κύριος Μισελ Κιχετά είναι ο Γάλλος συνάδελφος, ο συνάδελφος δηλαδή από το Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου ήταν πρόεδρος τμήματος ο κύριος Κιούμπικ είναι ο Πολωνός συνάδελφος από το Πολωνικό Ελεγκτικό Συνέδριο, ήταν και σύμβουλος του Προέδρου του Τμήματος και η κυρία Μπριγκίτε είναι η συνάδελφος από τη Λιθουανία και θα ήθελα να πω ότι η σημερινή συνεδρία θα πρέπει να θεωρηθεί προπαρασκευαστική. Θέλουμε δηλαδή μόνο να διερευνήσουμε και να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων για ενδεχόμενη θεσμοθέτηση τακτικών συναντήσεων μεταξύ ημών και ημών. Θα θέλαμε να σας ε, παρουσιάσουμε τα κύρια προβλήματα που επισημαίνουμε ως προς την ε, σύνδεση τη διασταυρωμένη την πολλαπλή συμμόρφωση και άλλα θέματα. Για να σας δώσω από την πλευρά μας δηλαδή τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει. Με την ε, άδειά σας λοιπόν κύριε Πρόεδρε θα λάβει το λόγο ο κύριος Κιούβικ και θα παρουσιάσει τις ε, διαπιστώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για την πολυπλησιμόρφωση και την αποσύνδεση και μετά θα θυμάστε βέβαια ότι ο κύριος Κρέτα είχε κάνει την παρουσίαση της ε, γνωμοδότησης για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠΑ πλευράς του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα σας ε, παρουσιάσει λοιπόν τα νέα στοιχεία για τις νέες προτάσεις μας για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. So I will start. Honorable members of parliament, ladies and gentlemen. Τιμή κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο κάνουμε τις διάφορες ε, ακροάσεις για την πολλαπλή συμμόρφωση, αυτό το οποίο κυρίως μας απασχολεί είναι τα κυρία θέματα που αφορούν την ΚΑΠ και κυρίως ποια είναι τα πιο τυπικά παραδοσιακά προβλήματα, αν θέλετε, τα οποία οι ελεγκτές μας βρίσκουν στον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ. Η μεγάλη πλειοψηφία των δαπανών αφορά τις άμεσες πληρωμές, νέσπιες και τα ΣΑΠΣ. Είναι λογική απόρρια των ε, πληρωμών αποσύνδεσης και κυρίως τρία θέματα θα ήθελα να τονίσω τα οποία βρίσκει και γράφει σε εκθέσεις της το Ελεκτικό Συνέδριο θέματα όχι σημαντικά για τις ε, κοινοτικέ καταβολές, αλλά κυρίως για την ε, φήμη την οποία στο σύνολό της έχει η ΚΑΠ. Πρώτα απ' όλα, οι δικαιούχοι, η πολλαπλή συμμόρφωση και οι διάφορα θέματα τα αποφορούν ε, την γη, την χρήση γης, ποιες είναι ε, κυρίως τα θέματα τα οποία φορούνται από τον ορισμό των ε, χορτολιβαδικών περιοχών. Πρώτα απ' όλα έχει σχέση αυτό με την επιφάνεια και το είδος ε, της ε, καλλιεργίας για να μπορέσει να είναι ε, να δικαιούται αυτό το κομμάτι γης ε, την ε, βοήθεια. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάποια χορτολιβαδική χώρη από κάποιες ε, χώρες θεωρούνται ως τέτοιες, ως ότι ε, δικαιούνται την ενίσχυση παρά το γεγονός ότι πολλές φορές πρόκειται για βραχώδεις περιοχές ή για δασικές. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει ε, στον εντοπισμό και στον ορισμό αυτών των χορτολιβαδικών εκτάσεων κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε, εάν δικαιούνται κάποια ενίσχυση, να τα ορίσουμε σωστά. Δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικό οι πληρωμές αποσύνδεση. Και εδώ, ποιος είναι ο ορισμός του αγρότη. Εδώ η κατάσταση και τα προβλήματα οφείλονται σε κάποιες αυσάφειες και στην ε, πολύ ευρία, ε, στον οποίο ευρύ ορισμό που δίδεται στον ε, αγρότη και στις δραστηριότητες του. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι κάποιες άμεσες καταβολές γίνονται σε άτομα τα οποία δεν ασχολούνται παρά μόνο πολύ περιθωριακά με αγροτικές ε, δραστηριότητες. Οι ενισχύσεις οι κοινοτικές για την υποστήριξη των αγροτών πολλές φορές, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνουν στις τσέπες μη αγροτών. Και στις δύο περιπτώσεις ε, το ελεγκτικό συνέδριο υποστηρίζει ότι θα πρέπει οι ενισχύσεις να γίνονται μόνον σε αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικοί αγρότες και ασχολούνται κυρίως με τις αγροτικές δραστηριότητες. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ποια είναι, ποιες είναι οι εκτάσεις οι οποίες ορίζονται ως χορτολιβαδικές και ποιες δικαιούνται και δικαιούνται την ενίσχυση και ποιοι είναι οι πραγματικοί αποδέκτες. Το το θέμα που θέλω να αναλύσω είναι το θέμα αυτό της πολλαπλής συμμόρφωσης. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της ΚΑΠ. Ίσως είναι το μοναδική αιτιολογία για τις άμεσες καταβολές, τις άμεσες πληρωμές. Αυτή η υποχρέωση πρέπει ε, να απορρέει από διάφορα ε, κριτήρια νομικού, νομικής φύσης τα οποία θα πρέπει να πληρώνται. Κάθε χρόνο στη συνέτησια έκθεση αναφέρουμε πολλές περιπτώσεις όπου δεν γίνονται ε, σεβαστές οι απαιτήσει αυτές. Κάποια τυπικά παραδείγματα είναι το ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες για την ευημερία των ζώων ή δεν πληρούν τα κριτήρια τα οποία αφορούν κάποιες καλλιέργειες. Θα πρέπει λοιπόν η πολλαπλή συμμόρφωση να είναι ως αρχή κάτι που ισχύει πάντα. Ως ε, συμπέρασμα θα πω ότι πολλές φορές δεν γίνονται οι σωστοί έλεγχοι και το σύστημα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο όπου εξαιτίας της πολυπλοκότητας δεν μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό συνιστούμε να απλοστευθούν και να διευκρινιστούν οι κανόνες και να δοθεί και, ιεραρχη, και ιεραρχικά προτεραιότητα στους κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να πληρώνται. Αυτές είναι οι συστάσεις που είχαμε κάνει στο παρελθόν και συνεχίζουμε να τις κάνουμε. Οι συστάσεις μας συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια την, ε, των ακρεώσεων που έγιναν και κατά τη διάρκεια αυτής της ε, νέας ε, οικονομικής κρίσης. Ο κύριος Κρετάνη θα σας προηγήσει περαιτέρω λεπτομέρειες του όλου συστήματος. Σας ευχαριστώ, περιμένω τις ερωτήσεις και θα σας απαντήσω. Mr. Chairman, honorable members, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα και μπορώ να σας μιλήσω σήμερα για τα όσα έχει πει στις εκθέσεις του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για τον έλεγχο που γίνεται στα πλαίσια της γεωργικής πολιτικής. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένε προποθέσει ελέγχου και επιλεξιμότητα, οι οποίε προποθέσει είναι κάπω πολύπλοκε. Επίση, βλέπουμε ότι γίνονται κάποιοι έλεγχοι προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι προϋποθέσεις αυτές τηρούνται. Πολλέ φορέ όμω δεν εφαρμόζονται σωστά οι έλεγχοι αυτοί, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι δαπάνε στην ανάπτυξη τη υπαίθρου ουσιαστικά μπορούν να οδηγήσουν πολύ συχνά σε σφάλματα. Όσον αφορά τώρα τους δικούς μας ελέγχου, εμείς προσπαθούμε να εξετάσουμε πραγματικά αν ε, οι ευρωπαϊκές επενδύσεις δημιουργούν μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Το βασικό ερώτημα είναι το εξή. Αν τα χρήματα έχουν δαπανηθεί σωστά ή αν καταφέρνει μέσω της χρηματοδότησης αυτής η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει τους στόχους της κατά τρόπο αποτελεσματικό οικονομικό. Βάσει διαφόρων ε, ελέγχων που γίνανε, σε πολλά μέτρα ανάπτυξη πέθρου τελευταία χρόνια, η απάντηση στο ερώτημα λοιπόν αυτό είναι η ακόλουθη, όχι, αρνητική απάντηση. Ο βασικός λόγος γι' αυτό είναι το ακόλουθο. Καταρχάς, ότι δεν έχουν εντοπιστεί ακριβώς οι ανάγκες και το ότι δεν έχουν ε, τεθεί σωστά οι στόχοι, δεν υπάρχουν οι σωστοί στόχοι στα πλαίσια τα μέτρα και υπάρχουν και στα πλαίσια των μέτρων και υπάρχουν κάποιες αδυναμίες όσον αφορά την παρακολούθηση, την εποπτεία. Θα αναφερθώ σε όλα αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία έχουν προγράμματα ανάπτυξη πέθρου, τα οποία δεν δικαιολογούν απόλυτα τις ανάγκες σε σχέση με τα μέτρα τα οποία έχουν επιλεχθεί. Και πολλές φορές έχουμε δει ότι οι στόχοι είναι πάρα πολύ γενικοί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να γνωρίζει κανείς ποιος είναι ο στόχος πίσω από τα μέτρα και επίσης ε, πώς μπορούμε τελικά να αξιολογήσουμε τα όσα έχουν επιτευχθεί μέσω των προγραμμάτων αυτών. Δεύτερον, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής δεν έχουν δημιουργηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιλέγονται τα καλύτερα δυνατά project, αυτά δηλαδή που αποκρίνονται στις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες των κρατών μελών και δεν κάνουν απαραίτητη διάκριση ανάμεσα σε καλά ή κακά σχέδια. Πολύ συχνά προσοχή έχει δοθεί απλώ στην δαπάνηση του κοινοτικού προπολογισμού, στη χρησιμοποίηση δηλαδή τη χρηματοδότηση, χωρί όμω να έχουν γίνει οι απαραίτητε επιλογέ. Αυτό ουσιαστικά θέτει εν κινδύνο και τον προπολογισμό της, ε, των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα, τον προπολογισμό των δικαιούχων. Επίση, δεν γίνεται επαρκή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων αυτών. Δεν είναι αξιόπιστη συστηματικά η αξιολόγηση αυτή και πολλοί δείκτε που έχουν χρησιμοποιηθεί δεν είναι κατάλληλοι δείκτε και οι έλεγχοι που έχουν γίνει από τα κράτη-μέλη όσον αφορά το value for money, δηλαδή έχουν αποδώσει οι χρηματοδοτήσεις αυτές δεν είναι πάρα πολύ καλοί. Γύρονται λοιπόν κάποια ερωτήματα για το τι τελικά επιτυγχάνεται μέσω της ευρωπαϊκής επένδυσης που γίνεται στην ανάπτυξη της υπαίθρου και το πώς ε, κάποιες ε, επιτροπές πολιτικές σαν τη δική σας μπορούν να ενημερωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα αποτελέσματα ή την επιτυχία ενός προγράμματος και πώς μπορούν ουσιαστικά πληροφορίες αυτές να διαμορφώσουν την μελλοντική πολιτική την οποία ακολουθούμε. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσοχή σας. Κύριος Κρέτα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Επιτροπή σας με κάλεσε πριν από μερικούς μήνες για να παρουσιάσω την ονότηση του Υπουργού Συνεδρίου για τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ για την νέα χρηματοδοτική περίοδο. Και χαίρομαι που είμαι σήμερα μαζί σας εδώ και για να μην επαναλάβω αυτά που είχα πει, θα αναλύσω τη γνωμοδότηση Επιτροπής βάσει των θέσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις συζητήσεις που έγιναν από τότε και εξακολουθούν βεβαίως. Ο ρόλος του συνεδρίου είναι να εξεταστεί η ε, σωστή δημονομική χρήση και να δούμε ποια είναι η σημασία την οποία προσδίδεται στην ΚΑΠ και στη χρηματοδότηση. Δυστυχώ, όσον αφορά τι άμεσε ενισχύσει, τα σχέδια κανονισμού που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναφέρουν τίποτε για τον στόχο των ενισχύσεων αυτών, είτε για τα αποτελέσματα που αναμένονται από την θέση εφαρμογή του. Αντίθετα με αυτό το οποίο είχε αναγγείλει η Επιτροπή και είχε διεκδικήσει, η νέα ΚΑΠ θα παραμείνει κυρίως μια πολιτική μέσων και όχι μία πολιτική με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων και ταυτοπίσιμων αποτελεσμάτων. Σήμερα η ΚΑΠ έχει τρεις αντικειμενικούς στόχους. Τον στόχο της παραγωγής, αύξηση της παραγωγής και της παραγωγία. Δεύτερον, υποστήριξη του ατομικού και επιμένου εισοδήματος του κάθε γεωργού. Πρόκειται για ένα από τους στόχους που περιλαμβάνεται συνθήκη και τρίτος στόχος, ο οποίος έχει μεγάλη σημασία παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ρητά στις συνθήκες, προστασία του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων όντων και του ζωικού βασιλείου. Και όπως είπε ο κύριος Κιούμπικ, αυτή η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος είναι σήμερα η μόνη αιτία, η αιτιολόγηση αν θέλετε, της καταβολής ενισχύσεως αγορούς. Πώς λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι στόχοι στη νέα ΚΑΠ. Η εξέταση του θέματος αυτός αποτελεί τον πυρήνα της γνωμοδότησης που δημοσίευσε το ελεγκτικό συνέδριο για τις νέες νομοθετικές προτάσεις. Για να μην μακρηγορήσω, θα αναφερθώ σε δύο από αυτούς τους στόχους. Την υποστήριξη στο εισόδημα και το πρασίνισμα της ΚΑΠ, του στόχο 2 και 3 μεταξύ αυτών που προανέφερα. Υποστήριξη των εισοδημάτων. Χωρίς διαμφισβήτηση, διαπιστώσαμε όλοι ότι συνεισέφερε η ΚΑΠ στην υποστήριξη αγροτικού εισοδήματος και στην ανατολική αισθητική πλευρά της Ευρώπης, αν θέλετε. Τι συμβαίνει όμως με το ατομικό εισόδημα που αναφέρουν οι συνθήκε. Δηλαδή τι γίνεται με την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των διαφόρων δικαιούχων. Δυστυχώς στο σημείο αυτό διαπιστώνεται ότι το πιο σημαντικό μέρος της ενίσχυσης, το 80% πηγαίνει στο, σε ένα μικρό αριθμό δικαιούχων, 20% ενώ η πλειοψηφία τους παίρνει μόνο ένα πολύ μικρό ποσό η πιο σημαντική ενίσχυση δίδεται στα υψηλότερα εισοδήματα και δεν νομίζω ότι αυτός ήταν ο στόχος ε, των ε, συντακτών της συνθήκες. Και, στην, ε, και παντού στην Ευρώπη έχουμε λοιπόν συγκέντρωση των ενισχύσεων προς αυτούς που έχουν τα υψηλότερα εισοδήματα και θα έλεγα ότι η συγκέντρωση είναι πιο σημαντική στην ανατολική πλευρά παρά στη δυτική της Ευρώπης. Και αυτό είναι άμεση απόρρινο συστήματος που βασίστηκε αποκλειστικά στις ε, ε, επιφάνειες προς εκμετάλλευση. Δεν υπάρχει λοιπόν στόχος όσον αφορά την κατανομή της ενίσχυσης. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα εδώ να κάνω τρεις παρατηρήσεις, τρεις διαπιστώσεις εκ μέρους μας. Πρώτα απ' όλα διαπιστώνουμε ότι κάποια στοιχεία της νέας νομοθεσίας τίνουν προς την ε, ε, επανισορρόπηση των εισοδημάτων των Δηλαδή, ε, η μη αναφορά των ιστορικών αναφορών σημαίνει ότι θα υπάρχει καλύτερη κατανομή μεταξύ των δικαιούχων. Επίσης, συμπληρωματική ενίσχυση ένα εκτάριο για τους νέους αγρότες. καθώς και η πρόταση που ψηφίστηκε από εσά για ενίσχυση ανά εκτάριο για τα πρώτα 50 εκτάρια της κάθε εκμετάλλευσης. Ή, τελευταία παρατήρηση, το συμπληρωματικό ποσό που ε, προβλέπεται για τους ε, αγρότες που ενεργούν με αντίξωες φυσικές συνθήκες. Όλα αυτά για να υπάρξει επανισορρόπηση της κατανομής των ενισχύσεων. Δεύτερη παρατήρηση. Διαπιστώνουμε ότι το Κοινοβούλιο, η δική σας Επιτροπή, ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για ανώτατο όριο των ποσών που δίδονται ατομικά ε, σε κάθε γεωργό. Αυτό το ανώτατο όριο τι σημαίνει. Από οικονομικής πλευράς δεν έχουμε πάρα πολύ ε, σημαντικές επιπτώσεις, αλλά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εδώ είχε λάβει εντελώς διαφορετική θέση. Δεδομένου ότι θέλει να γίνει το ανώτατο όριο αυτό να επιβληθεί και να οριστεί σε εθελούσια βάση από κάθε κράτος μέλος. Δηλαδή να αποφασίσει αν ναι ή όχι θέλει να ορίσει στις πιο υψηλές ενισχύσεις, τα μεγαλύτερα ποσά των ενισχύσεων, να επιβάλλει ανώτατο όριο. Και τελικά, τρίτο στοιχείο για την επανισορρόπηση, το ελεγκτικό συνέδριο, όπως είχε συστήσει, διαπίστωσε ότι οι ενισχύσεις μετά από τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής θα πήγαιναν στους ε, active farmers, σε αυτούς τους γεωργούς που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τις πραγματικούς αγρότες δηλαδή αν θέλετε. Πράγμα το οποίο θα επιλύσει και κάποια προβλήματα ε, κατανομής των ενισχύσεων. Ήταν πιο απλή η λύση που ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο απλή από αυτή της Επιτροπής, διότι πρότεινε τα κράτη-μέλη να κάνουν ονομαστικούς καταλόγους των ε, οντοτήτων που θα εξαιρούνταν από την καταβολή της ενίσχυσης αυτό είναι κάτι το οποίο είχαμε αναφέρει και σε πολλές προηγούμενες εκθέσεις μας, όπως Φερρυπίν, ε, δημόσια πάρκα στα κέντρα της πόλης, ε, ε, σιδηροδρομικές μενός, αεροδρόμια που δεν είναι η κύρια δραστηριότητά τους η γεωργία. Δεύτερη παρατήρωση και προσπαθώ να είμαι γρήγορος. Το πρασίνισμα της ΚΑΠ. Το πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα, όπως ξέρει, ε, έχει τρεις συνιστώσεις, καλύτερα από μένα. Τα λιβάδια, ε, η οικολογική ε, φυσική χώρη και οι εναλλακτικές καλλιέργειες σε χορτολιβαδικούς χώρους. Η καταβολή ενός συμπληρωματικού ποσού ανά εκτάριο προτείνουμε να γίνει παρά τα αποτελέσματα τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε. Στα κατεξοχήν και μονίμως ε, λιβάδια πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι δεν αλλάζει η επιφάνεια τους. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί όπως είπε και ο κύριος Κιούμπικ, η έννοια αυτή του μόνιμου λιβαδιού είναι κάτι το πολύ πλοκό να οριστεί με ευκρίνεια. Όσον αφορά την ε, μια εναλλακτικού τύπου καλλιέργεια. Ξέρουμε ότι αυτό το οποίο από οικολογικής πλευράς είναι σημαντικό είναι ε, τι γίνεται με τις εναλλακτικές καλλιέργειες για λόγους εφορίας. Όσον αφορά το τρίτο στοιχείο, τις οικολογικές ζώνες, τις προστατεύσιμες, ξέρουμε ότι είχε συμπεράνει το Συμβούλιο στις 6 και 7 Φεβρουαρίου και παραθέτω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ότι υπάρχει υποχρέωση να προβλεφθεί σε κάθε ε, αγροτική εκμετάλλευση ένας χώρος που θα θεωρείται ως οικολογικά ε, προστατεύσιμος χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στην, ε, στα έσοδα και στην εσοδιά του Γεωργού. Τελευταία παρατήρηση, πάντα για το πρασίνισμα της ΚΑΠ, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μία κάποια σύγχυση μεταξύ του πρασινίσματος για τον πρώτο πυλώνα και των ε, μέτρων των αγροτοπεριβαλλοντικών του δεύτερου πυλώνα. Στο δεύτερο πυλώνα, τα μέτρα που προβλέπονται επιτρέπουν χάρη του πρασινίσματος να καταβάλλονται κάποιες συμπληρωματικές ενισχύσεις. Δηλαδή, οι ίδιες πρακτικές που ισχύουν για το περιβάλλον θα καταβάλλονται δύο ε, φορές. Μία χάρη του πρώτου πυλώνα και μία χάρη του δεύτερου. Και εδώ είχε επικρίνει αυτό το κίνδυνο σύγχυση στο ελεγκτικό συνέδριο και επειδή θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός και διαφοροποίηση μεταξύ των δράσεων που επιβάλλονται σε όλους και καλύπτονται από την βασική ε, ενίσχυση που παρέχεται και Δεύτερον, κάποιων πιο απαιτητικών και ειδικών δράσεων που θα πρέπει να υποφελούνται από ειδική ενίσχυση στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον δεύτερο πυλώνα. Με τους νέους κανονισμούς πραγματικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση σύγχυσης μεταξύ των ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα και αυτών του δεύτερου πυλώνα. Και σταματώ εδώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Νομίζω ότι ε, οι παρεμβάσεις μπορούν να μας οδηγήσουν σε διάφορες σκέψεις αυτή τη στιγμή και βλέπω ότι στην αίθουσα είναι και οι συγητές μας οι οποίοι σε κάποια σημεία θα μπορούσαν να δώσουν κάποιες ε, διευκρινήσεις αυτό που ο κύριος κρετά για την ε, διπλή χρηματοδότηση. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στους αγορητές με τη σειρά που έχουν καταγραφεί. Μπορείτε να μου το πείτε βέβαια αν θέλετε να πάρετε το λόγο κι άλλοι. Άγνιου είναι ο πρώτος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν ζηλεύω τους, ε, τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου που έχουν να προσδιορίσουν τι σημαίνει χορτολιβαδική έκταση. Γιατί ύστερα από μια πολύ βροχερή μέρα μου έχει τύχει εμένα και στο δικό μου το χωράφι μάλιστα να έρθει η ελεγκτής και να μου πει εδώ πέρα δεν είναι χορτολιβαδική έκταση, είναι λίμνη. Αλλά ο ίδιος ελεγκτής μπορεί να πάει μετά σε μια ζεστή χώρα της Ευρώπης το καλοκαίρι και να δει μια και καυμένη ε, βουνοπλαγιά επειδή είναι καλοκαίρι και ο ήλιος καίει και να πει εδώ δεν υπάρχει χόρτο άρα δεν είναι χορτολιβαδική έκταση μόνιμα, μόνιμη. Άρα λοιπόν ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τον αγγλικό όρο parkland, γιατί όταν έχει κανείς 20 εκτάρια έκταση με ένα δέντρο, τότε γίνεται βέβαια απλό, απλά ορισμός ότι πρόκειται για μια χορτολιβαδική έκταση. Αλλά εάν υπάρχουν πολλά δέντρα, πώς θα ξεχωρίσουμε πού αρχίζει το δάσος και πού είναι χορτολιβαδική έκταση. Μην ξεχνάμε ότι στον ήλιο δίνει το δέντρο, την σκιά στα ζώα, δίνει το φρούτο, ενδεχομένως τον καρπό, δηλαδή και τα φύλλα που μπορεί να τρώνε. Και άρα θα πρέπει να είναι πολύ πιο σαφής ο προσδορισμός του πότε έχουμε να κάνουμε χρωτολιβαδική έκταση και πότε θα πούμε στον Γεωργό «Α, κύριε εδώ πέρα αυτό που έχεις είναι δασική έκταση και άρα δεν μπορείς να έχεις δικαίωμα σε ε, ενίσχυση». Επίσης ε, η εισαγωγή των διαφόρων ε, ε, ζυζανιοκτώνων και τα λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει πάρα πολύ την εικόνα του χορτολιβαδικού. Επίσης, τι είναι ο καλλιεργητής, τι είναι ο ε, γεωκτήμονας και πώς θέλει το ελεκτικό συνέδριο να επαληθεύσει ότι έχουν επενδυθεί χρήματα, έχει αναλάβει κάποιος ένα κίνδυνο επιχειρηματικό ή όχι, γιατί φαίνεται αυτές οι πληρωμές να πηγαίνουν στους γεωκτήμονες που όμως δεν έχουν κάνει καμία επένδυση και να έχουν αναλάβει κανένα κίνδυνο. Ευχαριστώ. Σικερίες και Μαγκίνες. και μετά Μαγκίνες. Κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι τέλεια η κοινή γεωργική πολιτική. Και μπορούμε να συμφωνήσουμε φαντάζομαι ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα. Ο τομέας εξαρτάται από από ειδικέ συνθήκες κλιματολογικές, γεωφυσικές και άλλες. Μια ποικιλία η οποία είναι ένα θετικό χαρακτηριστικό ασφαλώς της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και άρα νομίζω ότι είναι ε, υπερβολικό αυτό που ακούστηκε. Διότι βεβαίως πρέπει να είναι πιο ακριβείς οι ορισμοί για να τους εφαρμόζουν σωστά οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι. Αλλά όταν λέτε ότι δεν ε, είναι σαφές το τι κονδύλια έχουν πάει στη γεωργική ανάπτυξη κτλ. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να το πιστέψω. Έχουν παρουσιαστεί προτάσεις, έχουν αναλυθεί. Εγώ προσωπικώς έχω μιλήσει με τους γεωργούς πολλές φορές. Και διαπιστώνω ότι συχνά το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν είναι ενεργοί, δραστήριοι δηλαδή οι γεωργοί, αλλά ότι είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες από τη μια περιοχή στην άλλη. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά προβλήματα και πρέπει να προσέχουμε να μην αναλαμβάνουμε μέτρα τα οποία αποβαίνουν εις βάρος της γεωργίας μας. Αντί να λύνουμε τα προβλήματα. Ε, από τα λόγια σας φαίνεται σαν εννοείται ότι υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια των άλλων, αλλά δεν ισχύει αυτό. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρχουν κάποιε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι τόσο δεδομένο το πρόβλημα όσο νομίζετε. Μιλήσατε για εισοδήματα, ανταγωνισμό, προστασία του περιβάλλοντος, προαγωγή της υγείας. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί κανείς να θέλει μεγάλο εισόδημα, αλλά πρέπει να κοιτάμε και τον ανταγωνισμό. Και πρέπει να είμαστε βέβαιοι πάντοτε ότι κάθε εκτάριο είναι ανταγωνιστικό, παραγωγικό και Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μία ο, γνώμη, μια νέα μελέτη. Εκ τη δική σας, η οποία να φέρνει αντεπιχειρήματα, διότι φαίνεται να έχετε ενταχθεί μέσα σε ένα κύμα επικρίσεων εις βάρος της ΚΑΠ, που είναι πολύ, της, πολύ του σειρμού τώρα, ενώ όλοι εποφελούνται της ΚΑΠ. Ο μόνος, ο, αυτός που υποφελείται το λιγότερο στην τελευταία είναι ο ο Γεωργός. Μαγκίνες, παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συνεχίσω τα σχόλια του κυρίου Σερκέσκη για την ανάπτυξη της υπαίθρου και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η ανάπτυξη πέθρου είναι μια δύσκολη προσανάλυση πολιτική. Είναι πολύ δύσκολο να λύσουμε τις επιπτώσεις της. Ξέρετε ότι ε, εμπλέκονται διάφορες ομάδες ε, είτε σε προγράμματα κατάρτισης είτε σε άλλα προγράμματα και είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των προγραμμάτων αυτών. Θεωρώ ότι θα πρέπει όμως αυτή τη στιγμή να κρυβολογούμε λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω αν τα όσα μας είπατε είναι πάρα πολύ ακριβή σε σχέση με την πολιτική αυτή της ανάπτυξη πέθρου. Επίσης, αν ορισμένοι επιθυμούν αυτή την κατεύθυνση για την κοινή γεωργική πολιτική, δηλαδή περισσότερα προγράμματα ανάπτυξη πέθρου, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε και αυτά τα προγράμματα για την ανάπτυξη πέθρου. Φαντάζομαι όμω ότι των ζητημάτων αυτών θα πρέπει να επιληφθούν οι άνθρωποι που ασχολούνται πιο συγκεκριμένα με την ανάπτυξη πέθρου. Μια γενική παρατήρηση που θα έκανα. Ο κύριο Εκέρσκι μα είπε ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν είναι τέλεια. Μα τίποτα δεν είναι τέλειο, ούτε η επιστήμη είναι τέλεια. Εκτιμώ λοιπόν τις εκτιμήσεις οποίες κάνετε, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με την ανάλυση των παλαιών πολιτικών και την ίνερμηνία σας για το μέλλον. Νομίζω ότι όταν αναλύεται μια πολιτική είναι σημαντικό να εξηγείτε το γενικό της υπόβαθρο. Για παράδειγμα, όταν λέτε ότι 80% των πληρωμών πηγαίνουν σε ένα πολύ μικρό αριθμό δικαιούχων, τότε αυτό γίνεται ακριβώς επειδή η, το μέτρο αυτό η πολιτική συνεδεόταν με την παραγωγή. Άκουσα επίση ότι τα χρήματα πηγαίνουν σε αυτού που έχουν τα υψηλότερα εισοδήματα. Εγώ θα έλεγα προς το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ότι θεωρώ ότι άμεσες πληρωμές αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των εσόδων των αγροτών σε πάρα πολλά και χωρίς ενισχύσεις αυτές δεν θα είχαν κανένα απολύτως εισόδημα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η γνώμη του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά το ρόλο που τη δραματίζουν οι άμεσε ενισχύσει στην υποστήριξη του αγροτικού εισοδήματο. Θεωρώ ότι στι παρουσιάσει σα δεν ήσασταν πάρα πολύ ακριβής προς αυτό, σαφής προς αυτό. Επίσης ανησυχώ κάπως για το ακόλουθο. Το ότι είπατε ότι δίνουμε απλόχερα χρήματα σε πάρα πολλούς ανθρώπους και ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δικαιούχοι που παίρνουν το ίδιο, την ίδια οικονομική ενίσχυση χωρίς να καταλαβαίνουμε γιατί. Εφόσον το εισόδημα αποτελεί μέλος της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής θα πρέπει την αντίστοιχη ε, προσοχή να δίνουμε και στους υπόλοιπους στόχους, όπως η παραγωγικότητα για παράδειγμα. Έχετε για παράδειγμα αναλύσει το περιφερειακό σύστημα της ε, Γερμανίας, το οποίο είναι ένα μοντέλο το οποίο ακολουθεί την μονάδα αγροτεμαχίου που η ενίσχυση ουσιαστικά συνδέεται με το αγροτεμάχιο. Δεύτερη ερώτηση. Καθώ πηγαίνουμε προ μια πολιτική η οποία από ό,τι φαίνεται θα δίνει καταπο... κατακο... με συγχωρείτε πλέον, υποστήριξη ανεκτάριο, πολύ φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε στα, προβλήματα, στα, στα προβλήματα τα οποία έχετε εντοπίσει, ότι μεγάλοι γεωκτήμονες ουσιαστικά θα έχουν μεγαλύτερε ενισχύσει. Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπετε ότι πλησιάζουμε ακόμα περισσότερο στο ίδιο πρόβλημα, να το λύνουμε το πρόβλημα αυτό. Βλέπω επίσης ποια είναι η αποψή σας σε σχέση με τις προτάσεις που έχει ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω περαιτέρω ποια είναι τα σχόλιά σας και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι θα αναφερθούν στο ζήτημα των οροφών. Επίσης, αναφερθήκαμε στο ζήτημα της επιλεξιμότητας, της πολλαπλής συμμόρφωσης των δικαιούχων Ξέρω ότι αναφέρες, είπατε ότι δεν υπάρχει απλούστευση. Μα αναρωτιέμαι εγώ είναι ποτέ δυνατόν να απλουστεύσει κανείς τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης. Θέλω να ελπίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και στου επιτόπου ελέγχου. Αν όντω έχετε Εντελεχώ εξετάσει το ζήτημα αυτό, θα μπορούσατε σε μελλοντική σας έκθεση να μας πείτε πώς μπορούμε να πλουστεύσουμε το σύστημα της πολλαπλή συμμόρφωση. Ξέρω ότι στο παρελθόν έχω αναφερθεί προκλητικά στο ζήτημα αυτό, Πάντω θα ήθελα πραγματικά να γνωρίζω ποια είναι η δική σας άποψη. Να μας πείτε δηλαδή ότι ανακολουθώντα τα σημεία α, β, γ, Τις συστάσεις δηλαδή αυτές μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε την ε, πολιτική που ακολουθούμε. Γιατί τα σχόλιά σα ε, εν γέννη είναι καλά, αλλά είναι πολύ σημαντικό να επιφέρουν και μια βελτίωση. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του πρασινίσματο τη κοινή γεωργική πολιτική, το οποίο αναφερθήκατε, καθώς επίση και το ζήτημα τη βασική γραμμή πολιτική των διπλών πληρωμών και το καθεξής. Ξέρω ότι πολλέ φορέ ο τρόπο που είχε ψηφίσει για τα ζητήματα αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προκαλεί κάποια σύγχυση. Πάντω, στο δεύτερο πυλώνα υπάρχει μια βασική γραμμή η οποία βρίσκεται πάνω από το προσύνισμα. Και για του γεωργού που συμμετέχουν σε γεωργοπεριβολοντικά προγράμματα πέρα από το πρασίνισμα, θεωρώ ότι τα πράγματα εκεί πέρα βαίνουν αισίω και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αντίφαση στο να λαμβάνουν μια ενίσχυση για τη γεωργική του δραστηριότητα αλλά και για τις πρωτοβουλίες πρασινίσματος. Μάλλον εσείς δεν πρέπει να συμφωνείτε με αυτό. Κύριε Πρόεδρε, πολύ φοβάμαι ότι γίνονται πάρα πολλέ αναλύσει, αλλά δεν αναλύουμε παρκώ το τι ακριβώ θέλουμε να πετύχουμε, ποιο είναι ο τελικό στόχο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να καταλήξουμε αυτή τη στιγμή σε αποτελέσματα και όχι σε πηχαίου τίτλους στις εφημερίδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε προγράμματα αποτελεσματικά, τα οποία θα πρέπει να θεσπίζονται σε συνεργασία με του γεωργού. Και αν αυτό εσείς το εντοπίζετε ως διπλή χρηματοδότηση, τότε ας γίνει αυτό αποδεκτό εφόσον τα προγράμματα είναι θετικά. Και στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα μπορούμε να έχουμε και εταιρικέ σχέσει ευρωπαϊκέ για την κοινοτομία, όπου θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε του γεωργού να καταλάβουν ότι η κοινοτομία μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποφελή για την δική του την παραγωγή και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουν πραγματικά να προσαρμόσουν την παραγωγή τους στις νέες αυτές πρωτοβουλίες που μπορούμε να τους δώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συγκεκριμένε θετικές επιπτώσεις όσον αφορά την πρακτική που ακολουθείται επί τόπου, κατά την καλλιέργεια δηλαδή, είτε προέρχονται συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Αν θέλετε να βελτιώσετε πραγματικά την βιωσιμότητα, είτε πρόκειται για την παραγωγή, είτε πρόκειται για το εισόδημα, θα πρέπει από κοινού με του γεωργού να συνεργαστούμε, προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποιε πρακτικέ που θα είναι αποφελεί για αυτού. Οι δικέ σα προτάσει, για παράδειγμα, όσον αφορά την ε, αμυψισπορά, νομίζω ότι είναι σημαντικές, αλλά θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές και από τους ίδιους τους ε, γεωργούς. Ξέρετε ότι σε ορισμένε περιπτώσεις ε, έχετε ζητήσει ένα 10% από την γεωργική εκμετάλλευση να μην συμμετέχει πλέον στην παραγωγή. Πείτε το όμως αυτό στους ε, καταναλωτές, οι οποίοι ενδεχομένως να φοβούνται ότι οι τιμές κατά αυτόν τον τρόπο, οι τιμές των βασικών γεωργικών προϊόντων, ενδεχομένως να αυξηθούν. Επίσης, αν σε επίπεδο αγροκτήματος καταφέρνουμε να καταδείξουμε τα ωφέλη της ε, βιολογικής καλλιέργειας για τους ίδιους τους γεωργούς, για την ίδια την καλλιεργιά τους, ενδεχομένως να καταφέρουν τελικά να εγκρίνουν περισσότερα τέτοια μέτρα και να εφαρμόσουν τέτοιες γεωργικές μεθόδους. Επίσης, έχετε εντοπίσει κάποια σημεία, κύριε Κρετά, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά δεν τα έχετε αναπτύξει ιδιαίτερα κάποιες πληρωμές οι οποίες γίνονται για συγκεκριμένα αγροκτήματα, όπως επίσης και κάποιες άμεσες ενισχύσεις οι οποίες έχουν ως δικαιολόγηση μόνο την ευημερία των γεωργών. Ξέρετε ότι σε ορισμένε περιπτώσεις αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι κάποια εισοδήματα υπολείπονται πάρα πολύ από τα μέσα εισοδήματα που μπορούν να έχουν άλλε πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση αυτή θεωρώ ότι οι ενιαίε ενισχύσει είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Κάποιοι εκτινοτρόφοι, για παράδειγμα, ενδεχομένω να μην καταφέρνουν καν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά του αν δεν υπήρχαν οι άμεσε ενισχύσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν αυτέ οι άμεσε ενισχύσει για να έχουμε παραγωγή συγκεκριμένου τομεί, όπω για παράδειγμα παραγωγή βόλου Πολύ φοβάμαι πάντω ότι ορισμένα μηνύματα τα οποία στέλνονται προ τα έξω, ενδεχομένω από τα μάτια μαζική ενημέρωση, μπορούν να λειτουργήσουν πάρα πολύ αρνητικά σε σχέση με αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε εμεί ω Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι συστάσει τι οποίε δίνετε, αλλά με την άδειά σα πρέπει να σα πω ότι δεν είστε εκλεγμένα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί τελικά καλούμαστε να πληρώσουμε το τίμημα κάθε φορά που η κοινή γνώμη στρέφεται εναντίον μα ή εναντίον των συστάσεων που γίνονται εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω ότι εγώ είμαι πέρα από όλους υπόλογοι στην δική μου εκλογική περιφέρεια, ακριβώ επειδή οι άνθρωποι αυτοί με εκλέγουν. Και πρέπει να δικαιολογήσω κάποιε από τι προτάσει που κάνουμε στα πλαίσια τη κοινή γεωρική πολιτική. Ομολογώ ότι η μεταρρύθμιση τη κοινή γεωρική πολιτική αυτή τη φορά είναι η πιο δύσκολη, γιατί αυτό που θέλουμε είναι αποσυνδεδεμένε ενισχύσει, αλλά θέλουμε παράλληλα και υψηλή παραγωγή. Θέλουμε περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αλλά περιορίζουμε παράλληλα τον προπολογισμό. Αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και η πρόκληση είναι η ακόλουθη. Θα ήθελα πραγματικά το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο να μας πει τι θα γίνει με τις πληρωμές εκείνες οι οποίες συνδέονται με τα αγροτεμάχια. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία έχουν υιοθετήσει ενισχύσεις με βάση το εκτάριο. Ποιε είναι οι επιπτώσει έπειτα όσον αφορά τη γεωργία, την κτηνοτροφία. Τι γίνεται επίση με τι τιμέ των ίδιων των αγροτεμαχίων. Πολύ φοβάμαι ότι ενισχύοντα τι ενισχύσει, με το συνδέοντας με συγχωρείτε τι ενισχύσεις με το αγροτεμάχιο, ενδεχομένω να αυξάνουμε ιδιαίτερα τις τιμέ και ενδεχομένω να ενισχύουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πραγματικά γεωργοί. Διαβάζοντας τις εκθέσεις, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πραγμα ποιο είναι ο προσανατολισμό τον οποίο θέλετε να προωθήσετε όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, αλλά να μην επηρεαζόμαστε απλώ στην κριτική στι επικρίσει. Οι επικρίσει είναι απλώ επικρίσει και δεν μα οδηγούν αναγκαστικά σε έναν καλύτερο δρόμο, σε έναν πιο αποτελεσματικό προσανατολισμό. Κάθε φορά λοιπόν που κάνετε κάποιε επικρίσει, όταν λέτε ότι πρέπει να πλουστευτεί η πολλαπλή συμμόρφωση, πείτε μα πώ μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ. Τσαφεσκόφσκι και George Λάιν στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μετά από αυτά που η κυρία Μαγκίνη, κύριε Σαρκόφσκι, πριν από αυτόν, θα πω το εξή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και με ευχαρίστηση συμμετέχουμε σε αυτήν. Θα πάμε στο το εξής. Εκπλήσω με το, τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε αυτή τη τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου. Εγώ πρέπει να σας πω ότι στο παρελθόν ήμουν πρόεδρος του Πολωνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και ο γενικός κανόνας εθνικό επίπεδο είναι ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του πολιτικού σκέλους αν θέλετε και του ε, πραγματικού βάση των ορισμάτων στα οποία καταλήγει κάθε φορά το ελεκτικό συνέδριο και παίρνει κάποιες αποφάσεις. Σήμερα γίνονται διάφορες παρατηρήσεις που ξεπερνούν κατά κάποιο, ώρα, κατά κάποιο τρόπο τα όρια των αρμοδιοτήτων του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα ήθελα να έχω ακούσει κάποια συμπεράσματα μετά από τους ελέγχους που έγιναν. Έχω όμως την εντύπωση ότι δεν συμβαίνει αυτό σήμερα. Κάνουμε αλλά αναλύσεις των αποτελεσμάτων δεν έχουμε από ό,τι κατάλαβα μετά τους ελέγχους αυτούς διαπιστώσει ότι γίνονται πάρα πολύ μεγάλες ε, καταχρήσεις. Τουλάχιστον τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο στον τομέα των διορθωτικών ταμείων. Εγώ είμαι εισηγητής μιας έκθεσης για τα χρηματοπιστωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011 και έχουμε να κάνουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσά κατάχρησης των 77 εκατομμυρίων δις. Εδώ έχουμε να κάνουμε στην ΚΑΠ με μικρό ποσά. Ενώ το 40% των κονδυλίων του κοινοτικού προβλησμού πηγαίνουν στην ΚΑΠ. Άρα καταλαβαίνετε ότι αναλογικά δεν πρόκειται για μεγάλες καταχρήσεις και δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο κ. Κρετάν, δηλαδή ότι η μόνη αιτιολόγηση για την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Όχι, όχι, όχι. Η ασφάλεια των ειδών διατροφής είναι κατά την άποψή μου ο κύριος λόγος και η κύρια αιτιολογία, διότι η γεωργία στην Πολωνία δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την καταβολή άμεσων ενισχύσεων. Δεδομένου ότι οι μεγαλύτεροι ανταγωνισμοί μας στον πλανήτη μας ε, παίρνουν πάρα πολλές ενισχύσεις. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό θέμα για την ΚΑΠ. Και μην ξεχνάτε, υποστηρίζουμε τους αγρότες μας για να τρώμε ευρωπαϊκό ψωμί στην Ευρώπη. Και όχι για να αγοράζουμε το σιτάρι χωρίς καμία ασφάλεια αλλού ή πληρώνοντας σε προμηθευτές εκτός Ευρώπης κάποια ποσά πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεισφέρει στη συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά να μην κάνει πολιτικού περιεχομένου ε, ε αν θέλετε. Κύριε Λάιν, ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις. Έχω κάποιες ερωτήσεις μαζί με τους συναδέλφους. Ένα από, το θέμα, τα θέματα που πρέπει να λύσουμε είναι η, εσωτερική σύγκρουση στην ε, ΚΑΠ. Τι δηλαδή επιδιώκουμε με αυτήν. Άλλοι θεωρούν ότι αφορά την ενίσχυση του εισοδήματο. Οπότε, αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει, όπως συμβαίνει σε κάθε σύστημα πρόνοιας, να υπάρχει μια επαλήθευση ότι αυτός που λαμβάνει την ενίσχυση την αξίζει και όλα την ε, χρειάζεται. Οπότε με αυτή την περίπτωση μπαίνουμε σε πολλές δυσκολίες. Εγώ νομίζω ότι μπαίνουμε πέραν της απλής ενίσχυσης ε, εισοδήματος στην ε, προαγωγή δημόσιου αγαθού με δημόσιο χρήμα. Εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και με διαφορετικό τρόπο επαληθεύουμε το πώς αξιοποιούνται τα κονδύλια για το κοινό καλό. Άρα νομίζω ότι τίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να ε, κάνουμε και τις, σχετικ, τους σχετικούς, τις σχετικές προσαρμογές. Επίσης, ε, τα 2001 οι επιδοτήσεις ε, που δόθηκαν, ε, νομίζω ότι σωστά κατηγορούνται, ελέγχονται, αλλά από την άλλη είναι δύσκολο να αλλάξουμε από τη μια μέρα στην άλλη και δεν είναι και πολύ λογικό να ρίχνουμε χρήματα εκεί όπου δεν υπάρχει παραγωγή τροφής ή πολύ περιορισμένη παραγωγή τροφής. Και έτσι, όπως είπε και η Μαρή, πρέπει κάποιες από τις αλλαγές που είδαμε ήδη στη Βρετανία και την Γερμανία που εγκαταλείπουν το ιστορικό σύστημα και πάνε σαν σύστημα διαφορετικό πλέον, θα έπρεπε να επαληθευτούν και ενδεχομένω να εισαχθούν και αλλού. Αν και υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και αντιστάσει. Επίσης, μιλήστε για τον ενεργό λεγόμενο γεωργό. Υπάρχει ασφαλώς μια σειρά μέτρων που μπορούν να αξιοποιήσουν τα κράτη-μέλη για να ορίσουν ποιος είναι ενεργός γεωργός και ποιος όχι. Θεωρείται πάντως ότι μπορούν αυτά τα μέσα να βοηθήσουν την επαλήθευση ότι τα χρήματα που διατίθενται πάνε πράγματι σε αυτόν που ενεργά δραστηριοποιείται στη γεωργία και σε κάποιον που είναι αδρανής. Και η μετακύληση από τις άμεσες ενισχύσεις στην, περιφερειακή, στην ανάπτυξη πέθρου. Βλέπουμε ότι θα περιληφθεί στο κοινό πλαίσιο στρατηγικής η ανάπτυξη της υπαίθρου χωρίς ε, δίκτες παραγωγικότητας αλλά ούτε και ε, απορρόφησης. Αυτό λοιπόν ε, πώς βλέπετε να λειτουργεί. Και μια και αυτό θα ήταν για μένα χειρότερη λύση γιατί είναι πολύ περιπλοκά τα πράγματα το να προσπαθούμε δηλαδή να μετρήσουμε την απορρόφηση. Τώρα με ένα σύστημα στο οποίο εσείς στο ελεκτικό συνέδριο θα επαληθεύετε το, το εισερχόμενο, ε, θα σε επαληθεύσετε και το εξερχόμενο προϊόν. Ξανασυζητήσαμε και στο Λουξεμβούργο και θυμάμαι ότι κάποιος από εσά είχε ισχυριστεί ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβάρυνση κατά 40% του ελεκτικού καθήκοντος και φόρτου. Χρειάζεται πραγματικά τέτοιο. Δεν θα ήταν καλύτερο η Επιτροπή να καταλήψει την ιδέα της μέτρησης του εισερχομένου έναντι της επιλογής του εξερχομένου προϊόντος για να έχουμε μια καλύτερη λύση. Και να κοιτάμε μόνο τι παράγεται με βάση τους όρους του κοινοτικού πλαισίου. Ευχαριστώ. Κύριος Νίκολσον, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ χρήσιμη συνάντηση, γιατί με τι άλλο έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ανοιχτά και ειλικρινά. Πράγμα το οποίο λείπει. Καμιά φορά, έξω γι' αυτό αισθανόμαστε μια δυσφορία, γιατί αισθανόμαστε ότι αγωνιζόμαστε εδώ και όντω αγωνιζόμαστε. ξέρετε, εγώ έχω και 150 περίπου γεωργού στην ε, ε, περιφέρειά μου που δεν με αφήνουν σε χλωροκλαρί όταν πηγαίνω πίσω και πρέπει να τους εξηγήσω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα της γεωργίας. Εγώ δεν θα μπω στη συζήτηση το αν θα πρέπει εσείς να εμπλακείτε στον έλεγχο ή όχι. Τα έθιξαν οι άλλοι συνάδελφοι. Και καταλαβαίνω όταν λέτε ότι ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της υπαίθρου υπάρχει ανάγκη γιατί βλέπω προβλήματα και στη δική μου την περιφέρεια. Και έτσι διερωτώ με αν πράγματι τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα πάνε σωστά. Δεν υπήρχε καλύτερο τρόπο να αξιοποιηθούν. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, νομίζω, είναι αυτό. Και επίσης προσπαθούμε να φτιάξουμε μία λύση μονολυθική που να καλύπτει όλες τις περιφέρειες, όλες τις χώρες, ενώ ο καθένας έχει διαφορετικά προβλήματα στα οποία πρέπει να βρει λύσεις προσαρμοσμένες. Η δε ερμηνεία σε πολλές περιφέρειες που δίνεται στην κατάσταση οδηγεί σε συγκρούσεις συμφερόντων ακόμα. Συμφωνώ λοιπόν στην ιδέα μιας μεγαλύτερης ευελιξίας Αυτό είναι ο αγώνα μα Και με το επιχείρημα για το δεύτερο πυλώνα, για το πρασίνισμα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι το πρασίνισμα θα πρέπει να μείνει στο δεύτερο πυλώνα. Δεν έπρεπε να πάει στον πρώτο πυλώνα. Μόνο θα περιπλέξει τα πράγματα, θα καταστεί πιο δυσνόητο το σύστημα. Αυτό αντιμετωπίζουμε τώρα σαν πρόβλημα με τον πρώτο πυλώνα. Και στη τελευταία ανάλυση, πού είναι το όριο του πρασινίσματος υπό τον πρώτο πυλώνα και πού είναι το όριο σε σχέση με την ε, με το περισσότερο πρασινισμό του δεύτερου πυλώνα. Δυστυχώ δεν περιληφθεί η ευελιξία στην πρόταση αρχικά. Έτσι έχουμε βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση με προβλήματα. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, να βρούμε λύσεις. Δεν ρωτάμε θα είναι μια περιφέρεια κάνει σωστά, αν όχι. Σε αυτή λοιπόν τη φάση της μεταρρύθμισης Όλοι μιλάνε για λιγότερη γραφειοκρατία. Θα σας το πω ξεκάθαρα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε ότι αυτό που βλέπω τώρα εγώ, αλλά και από το πλευρά του Συμβουλίου, γιατί προσπαθούμε και εμείς να ολοκληρώσουμε τις, την επεξεργασία της θέσης μας και πάντα υπάρχουν τα προβλήματα, δεν συμφωνούν όλοι με το η θέση στην οποία καταλήγουμε και το Συμβούλιο προσπαθεί να καταλήξει μια θέση και μέχρι τέλους του μήνα θα πρέπει να ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Πώς θα συμφωνήσουμε δηλαδή. Ένα πράγμα που με απασχολεί όμω είναι το πώς θα προστατέψουμε, πώς θα εξασφαλίσουμε την επιβίωση των κοινωνιών, των κοινοτήτων της υπαίθρου. Από τη την εκλογική μου περιφέρεια βλέπω ξεκάθαρα ότι είναι όλο και λιγότεροι οι γεωργοί πλήρους απασχόλησης. Υπάρχουν κάποιοι που απασχολούνται μερικά στη γεωργία. Τώρα αυτό πώς μπορεί να εξασφαλίσει τη συνοχή της κοινωνίας, πώς μπορεί να εξασφαλίσει την παραμονή των σχολείων ή να μένουν ανοιχτέ οι εκκλησίες ή πώς θα αποτρέψει την διάλυση του κοινωνικού ιστού και, της ε, ανεργία, την ανεργία, δεν το έχουμε βρει ακόμα. Επίση, νομίζω ότι προσπαθούμε μερικές φορές να χρησιμοποιήσουμε τη γεωργική πολιτική ως υποκατάστατο μιας κοινωνικής πολιτικής για ορισμένες περιοχές της Υπέθρου. Ίσως θα καλό λοιπόν να κοιτάξουμε το πράγμα από άλλη σκοπιά. Αν και δεν νομίζω ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα το καταφέρει. Αλλά είναι αυτή η διαφορετική προσέγγιση ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να επιδιώξουμε. Όλο αυτό λοιπόν το θέμα, το πρασίνισμα, ο πρώτο πυλώνα, ο δεύτερο πυλώνα. Κοιτάξτε, κανεί δεν θέλει διπλή χρηματοδότηση. Κανεί ο σκανδαλοθυρικός τύπος έχει κολλήσει αυτό το θέμα τώρα. Γιατί είναι το μόνο το οποίο μπορούν να δουν και να καταγγείλουν με τη νέα ε, πολιτική, τη διπλή χρηματοδότηση. Αυτό εμείς θα πρέπει να το λύσουμε με το Δημήρη διάλογο και δεν νομίζω ότι θα πρέπει όταν καταλήξει αυτός να υπάρχει έστω και το, στο ελάχιστο η δυνατότητα της χρηματοδότησης. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Δηλαδή το να υπάρχει μια χρηματοδότηση μέχρι τα 50 εκτάρια και μετά επιπλέον, άνω των 50. Είναι διπλή χρηματοδότηση ή δεν είναι. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας δώσετε εσείς την ερμηνεία σας για το τι σημαίνει αυτή η χρηματοδότηση, αυτή η δυνατότητα χρηματοδότησης. Γιατί μένει με ανησυχεί αυτό. Έχω άλλωστε και διαρκή ε, διαρκείς επιθέσεις από τον τύπο και ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους αν είμαι υπέρ της διπλής ε, χρηματοδότησης των διπλών ενισχύσεων. Και η απάντηση φυσικά είναι αρνητική. Αλλά τελικά αυτό ο οποίο προσπαθεί και κάνει ευσυνήθειε προσπάθειε για την προστασία του περιβάλλοντο και, το, και τη οικολογία, τελικά βγαίνει χαμένο από αυτήν την ιστορία. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Και ίσως πρέπει και εσείς να αντιληφθείτε τι ε, εικόνα έχει ο ε, πολίτης. Αυτά που εμείς αντιλαμβανόμαστε από τις επαφές μαζί τους. Πρέπει να πω ότι περιμένω να, να είμαι σε θέση να πω στους πολίτες στην περιφέρεια μου ότι είδα κάτι εκπροσώπους του ελεγκτικού συνεδρίου και ότι τελικά θα μπορούσαμε να πείσουμε ότι δεν μπορεί κάποιος να κάθεται στο Λουξεμβούργο και να υπαγορεύεται τους ε, γεωργούς είτε στην ε, Ιρλανδία είτε στη Γαλλία είτε όπου αλλού ε, τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να κάνουν. Όχι, διότι ο Γιώργος δεν θέλει να κλέψει κανέναν. Ο Γιώργος θέλει να δουλέψει μέσα στο σύστημα με καλούς όρους, με σωστούς όρους. E Ευχαριστώ, Μάρτιν. Χόισλινγκ και μετά η Λουίζ. Ναι, έχουν καρφεί τα περισσότερα θέματα. Η πρόταση σας για τακτικό, σε τακτά διαστήματα δηλαδή διάλογο, είναι ευπρόσδεκτη ασφαλώς. Αλλά φαντάζομαι ότι θα συνομιλείτε και με το Συμβούλιο Γεωργίας Τουλάχιστον αυτό αναμένω να συμβαίνει. Και έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες στα θέματα αυτά. Αυτά τα οποία θίξατε στην αρχή των παρεμβασιών μας, παρεμβασιώσασταν ήταν αυτά τα οποία και μας μας έχουν απασχολήσει από την αρχή. Ο ενεργός ή δραστήριος γεωργός, σε παραδείγματι, είναι ένα θέμα στο οποίο έχει επιτευχθεί ευρεία συνένεση αυτό αφορά τη Γερμανία φυσικά, αλλά ίσως και άλλα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ε, κάποιοι γεωργοί, αρκετοί γεωργοί μερικής απασχόλησης που συμπληρωματικά μόνο ε, ζουν από την γεωργία, συμπληρώνουν μόνο το εισόδημά τους δηλαδή από τη γεωργία, αλλά, αλλά μπορεί να παίρνουν και τις σχετικές ενισχύσεις. Δεν θα έπρεπε τότε να μιλήσουμε για εισόδημα. Δεν θα έπρεπε αυτοί οι οποίοι αποφελούνται από τις ρυθμίσεις να βγουν έξω από το σύστημα. Από την άλλη, η κερδοσκοπία κάποιων επιχειρήσεων που επενδύουν στη γεωργία, κεφάλαιο, για τεράστιες εκτάσεις, στις οποίες όμως δεν υπάρχει γεωργός. Έχετε σε αυτό το θέμα κάποια απάντηση. Θα ήθελα να συζητήσουμε αν είναι δυνατόν. Ένα άλλο θέμα που ασχολούσε τον κύριο Λάνιν ήταν ε, αυτό των χορτολιβαδικών εκτάσεων. Το permanent pasture, μόνιμη χορτολιβαδική έκταση, είναι νομίζω η καλύτερη λύση, ο καλύτερος ορισμός. Γιατί ο όρος ε, λιβάδι, ε, η παιδιάδα δεν ε, σημαίνει απαραίτητο ότι υπάρχει χορτάρι. Και ότι μπορεί να βοσκήσει το ζώο εκεί αν πάμε από την άλλη στην Αυστρία, το Τυρόλο, ε, σε ορεινές περιοχές δεν είναι δυνατόν να κάτσει κανείς να μετράει το κάθε λιθαράκι για να το αφαιρέσει από τη συνολική έκταση προκειμένου να βρει ποια είναι η καθαρή χορτολιβαδική. Όμως κάπως πρέπει να βρούμε μια λύση και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε μια λύση για να στηρίξουμε αυτές τις περιοχές, αυτές τις ζώνες, ώστε να μπορεί και να συνεχίσει εκεί να ζει ο κτηνοτρόφος εν προκειμένου. Και επίσης υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπως στη Γερμανία, εκτατικές καλλιέργειες, οι οποίες μπορεί πλέον να μην έχουν να δώσουν μεγάλα νούμερα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη χρησιμότητα οικολογική. Επίσης αναφερθήκατε στο δεύτερο πυλώνα και τα γεωργικά τα μέτρα για την προχωρή της γεωργίας. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δούμε το θέμα της αξιολόγησης των μέτρων, πέραν των μέτρων των ίδιων. Δηλαδή, εάν υπαχθώ σε ένα πρόγραμμα ε, θα πρέπει μέσα σε ένα-δύο χρόνια να είμαι σε θέση και να ε, αποδείξω ότι έφερε αποτέλεσμα για, την, ε, για το περιβάλλον, ότι ήταν ωφέλιμο για το περιβάλλον. Σε ένα άλλο θέμα στην ενίσχυση με μέχρι 100 ευρώ στο εκτάριο δεν νομίζω ότι κάνει κανείς άλματα, δεν κάνει ουσιαστική πολιτική, μόνο συμπληρωματική βοήθεια μπορεί να προσφέρει. Και για τους στόχους της ΚΑΠ πολιτικά μόνο μπορούμε να τους κρίνουμε, πολιτική στοχή είναι, είναι μια πολιτική, ένα πολιτικό δίλημα το οποίο θα πρέπει να κρίνουμε με τους τρεις κύριους στόχους και τις προτεραιότητες που θα θέσουμε. Ναι, μπορεί να επιτυγχάνονται κατά σε διαφορετικό βαθμό, αλλά αυτό εξαρτάται σε, ένα βαθμό και από τα κράτη, πώς θα αξιολογήσουν δηλαδή την απόδοση αυτών των στόχων και των μέτρων. κράτη με μικρή έκταση έχουν ακόμη μεγαλύτερες ε, ε, ανισορροπίες ως προς τις πληρωμές. και δεν μπορεί να γίνει διόρθωση αυτών των ανισοτήτων ακόμη και αν δώσουμε τριπλάσια ενίσχυση στο γεωργό των κρατών αυτών. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στις προδιαγραφές ελέγχου στα κράτη-μέλη. Τις αξιολογήσατε. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να πούμε ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα διαφορετικό σε διάφορα μέρη του, ευρωπαϊκό σύστημα με διαφορετική ε, εικόνα σε διάφορες περιφέρειες ή ε, προτιμούμε να πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα ενιαίο σύστημα και αναλόγως να κάνουμε παληθεύσεις ε, ποιότητας κατά περίπτωση. Ευχαριστώ Λουίς και μετά ο Πέτερ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες του ελεγκτικού συνεδρίου για τις ε, απόψεις τους. Μου αρέσει να ακούω όλων τις απόψεις. Με κάποιες συμφωνώ και με άλλες δεν συμφωνώ βεβαίως. Αλλά αυτό είναι απόρρια της ε, πολιτικής συζήτησης και νομίζω ότι είναι καλή η ανταλλαγή απόψεων που κάνουμε με τους συναδέλφους. Πολλές ε, παρατηρήσεις είχαν πραγματικά πολιτική απόχρωση. Και ίσως αυτό έγινε για να μας βοηθήσει να νομοθετήσουμε καλύτερα. Κάποια σύγχυση όμως δημιουργήθηκε, διότι ο διαχωρισμός των εξουσιών εδώ δεν είναι απόλυτα σαφής. Οι βουλευτές πρέπει να νομοθετούν και τα δικαστήρια πρέπει να εφαρμόζουν τις πολιτικές αποφάσεις. Γι' αυτό κάποιες συστάσεις νομίζω ότι ξεπέρασαν το ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου και ελπίζω ότι κάποια μέρα θα μπορέσουμε και εμείς να έρθουμε στο ελεγκτικό συνέδριο και να πούμε και εμείς τη γνώμη μας για τον τρόπο με τον οποίο εσείς λειτουργείτε, να κάνουμε και εμείς επικρίσεις για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς τον πρόεδρο και τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου να διορθώσουν ενδεχομένω κάποια από τα σφάλματα που διαπράττουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ για τη συζήτηση. Όταν έχουμε εντατικό διάλογο με το ελεκτικό συνέδριο, Βεβαίω, και θέλω να ακούω πάντα επικρίσεις. Εγώ είμαι από αυτούς που, δεν, ε, που χαίρονται να ακούνε επικρίσεις. Γιατί πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και το βαθμό της αποδοχής των μέτρων. Έχει λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο και μια ματιά ως προς την αποδοχή των νομοθετικών μέτρων και έτσι είμαστε σε θέση να κάνουμε και μια δίκαιη, ισότιμη, τίμια συζήτηση ε, για το τι ισχύει και τι προκύπτει από τα μέτρα. Αλλά με μια προκατακτική ε, παρατήρηση θα ήθελα να πω ότι η πολιτική της Γεωργίας είναι και μια πολιτική ασφάλειας η οποία έχει τίμημα. Ή αλλιώς εγκαταλείπουμε το στόχο της ασφάλειας. Αν πούμε θα μπορούσε να γίνει συζήτηση. Ότι δεν μα ενδιαφέρει ποιο στόχο τη ασφάλεια, τον εγκαταλείπουμε. Άλλη μια προκατακτική παρατήρηση για τι άμεσε ενισχύσει. Παρακολουθώ από το 92 την κατάσταση και έχω αντιληφθεί ότι με τη διαμόρφωση των αμεσών ενισχύσεων, ε, την πολλαπλησή μόρφωση, την αποδέσμευση, προσπαθούμε να καθιδρήσουμε μια επιχειρηματική γεωργική δραστηριότητα. Αλλά από την άλλη πρέπει και να ικανοποιήσουμε την, τον όρο της ασφάλειας, δηλαδή επαρκή προμήθεια τροφίμων για τους πολίτες. Άρα Πρέπει να έχουμε την δυνατότητα της ετήρησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με την παραγωγή και ταυτόχρονα ένα ικανοποιητικό εισόδημα για τη γεωργική επιχείρηση, εκμετάλλευση. Εάν οι τιμές είναι καλύτερες ε, στις αγορές, ε, μπορούμε να μειώνουμε τις άμεσες ενισχύσεις. Αυτό θα ήταν ο όρος, φαντάζομαι. Και αν κοιτάξουμε λίγο τους πίνακες που δίνουν τη χρονική γραμμή, μειώνονται ε, από το 92 μέχρι τώρα οι άμεσες ενισχύσει. Άρα κάτι έχει καταλάβει και η ε, επιχειρηματική αυτή γεωργία, όπως επισημαίνει το ελεκτικό συνέδριο, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Και τώρα περνώ σε μια άλλη παρατήρηση, ότι προέρχομαι από μια περιοχή που έχει μεγάλες σχετικές ε, επιχειρήσεις, 20% των επιχειρήσεων έχουν το 80% των ε, ενισχύσεων από τον πρώτο πυλώνα. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι όποιος παίρνει την ε, ε, ενίσχυση για τα 10 εκτάρια μπορεί να την πάρει όπως είναι, αν κάποιος έχει μεγαλύτερη έκταση τότε παίρνει μόνο ένα ποσοστό. Αλλά από την άλλη είναι τόσο περίπλοκη κατάσταση θα μπορούσαμε να πούμε ότι βγάζουμε από το σύστημα όλες τις, όλες εκμεταλλεύσεις που είναι πάνω από 50 εκτάρια έκταση 5.000 εκτάρια οπότε βλέπουμε μόνο, στρεφόμαστε μόνο προς τις πιο αδύναμες οικονομικά εκμεταλλεύσεις και στηρίζουμε μόνο αυτές. 5.000 ευρώ λέει τώρα ο μιλητής. Ο μιλητής. Οπότε κοιτάμε τις ε, μικρότερες και πιο αδύναμες οικονομικά εκμεταλλεύσεις. Μια άλλη αλλά πρέπει αυτό το, το σκεπτικό να το πάμε μέχρι τέλους και να πούμε σε μια δεύτερη ανάγνωση ότι ε, εγκαταλείπουμε την άμεση ενίσχυση ανά επιχείρηση. Απλό. 3.000 ευρώ, το χρόνο σημειώνω έτσι, είναι εφάπαξ καταβολή, τα διαγράφουμε. Το θέλουμε όμως αυτό. Και τρίτο, για το κάπινγκ ή ε, για άλλε λύσεις που θα μπορούσαν να μας απαλλάξουν από πολλά προβλήματα. Γιατί ούτε εδώ έχει κηρυχθεί τίποτα ακόμα. Πέραν μιας ε, πολιτικής ερμηνείας, ενδεχομένω. Επομένως, ε, εγώ δεν θέλω από τη μια να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε επιχειρήσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή με τη μορφή της επιχειρήσεως, αλλά όταν έρθει η ώρα να τη στηρίξουμε να μην έχουμε το θάρρος και την παρεσία. Και τρίτον, υπάρχουν σφάλματα, έχουν εντοπιστεί σφάλματα. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το ότι ε, προσπαθούμε να χαράξουμε μια πολιτική από τη βάση προς τα άνω και όχι από τα άνω προς τα κάτω. Βέβαια τώρα φαίνεται η πολιτική να χαράζεται από τις Βρυξέλλε και να επιβάλλεται. Άρα η συμμετοχή των περιφερειών των μικρότερου, του, του μικρότερου επίπεδου με τις πρωτοβουλίες που μπορούν να αναπτύξουν γιατί μπορούν αυτές οι πρωτοβουλίες να προξενήσουν κάποια λάθη, αλλά χρειάζεται να συμμετάσχουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Βέβαια εδώ χρειάζεται να δείξουμε κατανόηση πέραν της περίπτωσης στην οποία διαπιστώνεται απάτη. Αλλά μικροσφάλματα μπορούμε να κάνουμε δεκτά. Για τη διπλή ενίσχυση, η στήριξη. Εδώ μπορούμε να είμαστε πολύ επικριτικοί, όπως άλλωστε είδαμε και με, την, με το δεύτερο πυλώνα για το, πράσινο, για το πρασίνισμα, για το εξορισμό πρασίνισμα, όπου πρέπει να πούμε ότι είτε δεν επιτρέπουμε τη διπλή ενίσχυση για καμία γεωργική εκμετάλλευση, είτε πρόκειται για οικολογική, είτε πρόκειται για συμβατική ε, γαλλιέργεια, ή αλλιώς ε, το υπεριορίσουμε μόνο σε όσες έχουν περιβαλλοντικά προγράμματα, ειδικά περιβαλλοντικά προγράμματα. Ευχαριστώ. σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ο κύριος Σαρμάς έχει τώρα το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να πω με τη σειρά μου ότι οι συζητήσεις αυτές είναι πάντα ιδιαίτερα επικοδομητικές. Μας επιτρέπουν να καταλάβουμε καλύτερα ο ημέν τους δε. Όχι επειδή εμεί θέλουμε να σπρώξουμε το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο να κάνει μια διαφορετική δουλειά από αυτή την οποία κάνει, να κάνει κάτι διαφορετικό από τις αρμοδιότητές του. Εννοείται ότι ε, η πολιτική ευθύνη είναι η δική μας. Ε, είναι δική μας. Εμείς είμαστε νομοθέτες, εμείς και το Συμβούλιο. Θεωρώ πάντως ότι οι αξιολογήσεις του Ευρωπαϊκού Λεκτικού Συνεδρίου μπορούν να μας βοηθήσουν να νομοθετήσουμε καλύτερα, να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα τα οποία λογικά αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια μιας τόσο πολύπλοκης νομοθεσίας όπως είναι η κοινή γεωργική πολιτική. Θεωρώ ωστόσο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα σε σχέση με την ψηφοφορία την οποία είχαμε στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινήθηκε προς μια θετική κατεύθυνση. Αν θυμάμαι τουλάχιστον ε, καλά, όταν είχαμε μαζί μας τον κύριο Κρετά εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε αναφερθεί στο ζήτημα αυτό, στην κατεύθυνση που έπρεπε να πάρει κοινή γεωργική πολιτική. Ε, μπορώ να δώσω τώρα αυτή αμέσω το λόγο στον κύριο Ιωάννη Σαρμά για την πρώτη απάντηση και έπειτα μπορείτε να, να αποφασίσετε εσεί ποια σειρά θα ακολουθήσετε στι υπόλοιπε απαντήσει οποίε θα δώσετε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διαθεσιμότητά σα που είστε εδώ και μπορείτε να απαντήσετε. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήραν το λόγο. Μας θέσανε ερωτήσει και κατάφεραν να εκφράσουν επίση τη δική του την άποψη. Πρωτού πάρουν το λόγο συναδελφοί μου για να απαντήσουν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που ετέθησαν, θα ήθελα να διευκρινίσω δύο πράγματα εκ των προτέρων, για να αποσαφηνίσω μια παρανόηση που έχει γίνει ενδεχομένω. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο έχει δύο αρμοδιότητες βασικές. Η πρώτη είναι να υποβάλει ελεκτικές εκθέσεις και η δεύτερη είναι να γνωμοδοτεί επί των νομοθετικών σχεδίων που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των οικονομικών των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο ευρωβουλευτές που πήραν όμως το λόγο, συγγνώμη, δύο συνάδελφοί μου οι οποίοι πήραν το λόγο, σας παρουσίασαν το περιεχόμενο δύο ελεγκτικών εκθέσεων λοιπόν με τις παρεμβάσεις αυτές, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι οι παρεμβάσεις αυτές, οι εκθέσεις αυτές βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, σε πράγματα τα οποία απευθύνονται ή παραβιάζονται συγκεκριμένα ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα πρέπει να τηρούνται στο σύστημα πληρωμών και ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις ελεγκτικές εκθέσεις θεωρώ ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Προφανώς μπορούν να υποβληθούν κάποιες ε, επικρίσεις. Όπως σας είπα, υπάρχουν και κάποιες άλλες αρμοδιότητες οποίες έχουμε, συγκεκριμένα να μπορούμε να γνωμοδοτούμε για νομοθετικά σχέδια, για σχέδια νομοθετικών πράξεων. Προφανώς εμείς λειτουργούμε ως Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνεδρίο, αλλά οι εκθέσεις αυτές δεν είναι ελεκτικέ εκθέσει, εκθέσεις, είναι μία γνώμη, μία γνωμοδότηση για ένα νομοθετικό κείμενο. Βεβαίω και στην περίπτωση αυτή εμείς λειτουργούμε ως οργανισμός επαγγελματιών, τεχνοκρατών και όχι ως πολιτικός οργανισμός. Οι γνωμοδοτήσεις μας λοιπόν για τα νομοθετικά κείμενα στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Κρετά βασίζονται είτε στην εμπειρία την οποία διαθέτουμε από το παρελθόν, δηλαδή κάθε φορά που εντοπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, η οποία προτείνει ένα κείμενο, επιθυμεί να διατηρήσει τελικά ένα κείμενο το οποίο δημιούργησε εν τέλει προβλήματα, τότε εμεί επεμβαίνουμε και ουσιαστικά υποβάλλουμε μία γνώμη. Λέμε ότι κοιτάξτε, δεν λάβατε υπόψη στην πρόταση την οποία κάνατε τις δικές μας τις προτάσεις, τις δικές μας παρατηρήσεις. Επίσης επεμβαίνουμε όταν εντοπίζουμε στα πλαίσια νομοθετικών κειμένων αντιφατικούς στόχους ή αν βλέπουμε ότι τα μέσα τα οποία προβλέπονται δεν αρκούν για να επιτευχθούν οι στόχοι. Πέραν από όλα αυτά, ουδέποτε κάναμε κάποια πολιτική τοποθέτηση για νομοθετικό κείμενο. Ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο. Αρμοδιότητά μας, όπως εξήγησε, είναι να υποβάλουμε μια γνωμοδότηση, να καταθέσουμε μια γνωμοδότηση όχι ως ελεγκτές, μια γνωμοδότηση για ένα νομοθετικό κείμενο, για ένα σχέδιο, νομοθετικό κειμένου, για ένα σχέδιο νομοθετικού κειμένου βάσει πάντα επαγγελματικών τεχνικών κριτηρίων. Η δεύτερη παρατήρηση με την άδειά σα, κύριε Πρόεδρε, η δεύτερη διευκρίνηση, αποσαφήνιση αν θέλετε, είναι η ακόλουθη. Είδαμε για παράδειγμα ότι έχουν ε, εντοπιστεί κάποια προβλήματα όσον αφορά τους βοσκοτόπους και, τις ε, σχετικές, και τους σχετικούς ελέγχους. Δεν καθορίζουμε εμεί τους κανόνες ελέγχου όμως. Οι κανόνες αυτοί υφίστανται και εμείς καλούμεθα να τους ερμηνεύσουμε. Αυτό το οποίο μπορεί να μας προσάψετε είναι ότι δεν ερμηνεύουμε σωστά το κείμενο. Δεν είναι πάντως το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο το οποίο θεσπίζει τους κανόνες το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ερμηνεύει τη σωστή εφαρμογή των κανόνων και θεωρώ ότι αυτό το κάνουμε με έναν σίγουρο ρεαλισμό, με έναν βέβαιο ρεαλισμό. Και προσπαθούμε να δείξουμε την καλύτερη δυνατή κατανόηση, αν θέλετε, των κανόνων αυτών, την καλύτερη δυνατή ερμηνεία. Αν λοιπόν οι επικρίσει έχουν να κάνουν με του κανόνε αυτού καθ' αυτού, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο δεν θεσπίζει του κανόνε, αλλά προσπαθεί να του ερμηνεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ελέγξει αν εφαρμόζονται οι κανόνε αυτοί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήθελα να δώσω καταρχά το, το λόγο στον κύριο Κιούμπικ, στη συνέχεια στην κυρία Μπαντμπερίτε και στη συνέχεια στον κύριο Κρετά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω τις ερωτήσεις των Πολωνών συναδέλφων, Τσοκέρσκι και Βοσκόφσκι. Και θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Ο διαχωρισμός αυτός είναι η, η πραγματικότητα των ρόλων μας είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα και στο τέλος αυτής της νέας περίοδου, της νέας περίοδου των δημοσιονομικών προοπτικών παρουσιάζουμε τις θέσεις μας ε, στοιχειοθετημένες, στι, ε, εμπεριστατωμένες και μας επισημαίνεται ότι εμείς επιδεινώνουμε τις, ε, τις ε, υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα στις καταχρήσεις και τις απάτες. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εμείς επισημαίνουμε την απουσία σεβασμού των ε, κανόνων και το πρόβλημα της ανυπαρξίας ορισμένων ε, ορισμών ως προς τις γέες και ως προς τους γεωργούς. Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται αυτοί οι ορισμοί να προσδιοριστούν τόσο ως προς τις γέσεις ως προς το Γεωργό και δεν θέλω να πω ότι όντως μπορεί να υπάρχουν κάποιες ε, παρατυπίες. Ο κύριος Σικέρσκι μιλάει για 5% παρατυπίων στην ΚΑΠ. Ναι, η ανάλυση ε, των ε, DAS τα τελευταία χρόνια αυτό μας δείχνει. Αλλά ο κύριος Σικέρσκι θεωρεί ότι η δική μας τοποθέτηση είναι, αποβαίνει εις βάρος της ΠΑΚ, ότι είναι αντίθετη με τους στόχους της ΠΑΚ. Δεν είναι αλήθεια όμως αυτό. Εμείς προσπαθούμε μόνο να βελτιώσουμε την ΚΑΠ και την εφαρμογή των κανόνων της. Εμείς προσπαθούμε να θέσουμε αυτή την ε, πολιτική, την ΚΑΠ, στην υπηρεσία των ε, πολιτών. Ευχαριστούμε. Έχουμε περιθώριο μέχρι τις 6 και 40. Παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο σας και έχετε το λόγο. Θα σου το τηλέφωνο. I'd like to speak on rural development. Θα ήθελα να μιλήσω για θέματα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Ρωτήσατε πώς μπορούμε να δαπανούμε έξυπνα και πώς μπορούμε σωστά να κάνουμε εκτίμηση των δαπανών για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Κάνουμε τη σωστή αξιολόγηση. Σωστό είναι αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι και για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε την αξιολόγηση της ε, απόδοσης των κονδυλίων που καταβάλλονται και των επιπτώσεων των δαπανών για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Πρέπει όμως να πω ότι υπάρχουν οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίζονται στους κανονισμούς, αλλά δυστυχώς πολλές φορές κατά τη δική μας ερμηνεία είναι κάποιοι ε, κανόνες πάρα πολύ γενικόλογοι και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν για τις ειδικέ ανάγκες και όλες αυτές οι ανάγκες να εκφράζονται με σαφήνεια όσον αφορά τους στόχους και την στόχευση για την ε, επίλυσή τους. Και υπάρχει και διακριτική ευχαίρεια βεβαίως ε, των ε, κρατών μελών για τις ανάγκες, για την υλοποίησή τους και για τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουν. Και αυτοί αποφασίζουν ποια είναι τα κριτήρια και οι κανόνες επιλεξιμότητας. Και όταν κάνουμε εμείς ε, τις διάφορες ε, ακροάσεις και τους ελέγχους Φερρυπίν, για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις βλέπουμε ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά τις ανάγκες και τον τρόπο με τον οποίο θα ικανοποιηθούν. Άλλοι όμως όχι. Εξάλλου, όταν ε, ε, έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου, δεν έκανε στοχοθέτηση των μέτρων με σαφήνεια. Εάν θέλετε να υλοποιήσετε κάποιους στόχους, πρέπει πραγματικά να το κάνετε βάσει ενός πολύ ακριβόλογου συστήματος. Όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, θα πω ότι τα μισά χρήματα δαπανώνται για σχέδια επενδύσεων. Σχέδια επενδύσεων. Τι σημαίνει. Ε, δημόσιες προμήθειες, πολύ καλό προγραμματισμό, εμπλοκή του δημοσίου και υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις κρατικές προμήθειες. Και πάντα συνιστούμε να γίνει απλοποίηση των, κανόνες, των κανόνων αλλά να έχουμε και ένα σαφές σύστημα στοχοποίησης των στόχων. Παρακαλώ να συντομεύσετε, λέει ο Προεδρεύων. Τελείωσα, τελείωσα, λέει η ομιλήτρια. Πολύ καλά. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο-τρεις ερωτήσεις. Το θέμα των, θέμα των στόχων που τέθηκε από τον κύριο Άγνιο, από τον κύριο Λάιον και εν μέρει από την κυρία Μαγκίνες. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν καθορίζει τους ε, στόχους της ΚΑΠ. Αυτό το οποίο επικρίνουμε εμείς ε, είναι η έλλειψη στόχων. Εάν διαβάσετε το Γενικό Κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις και βρείτε πού αναφέρονται οι αντικειμενικοί στόχοι της ΚΑΠ, θα σας είμαι ευγνώμων, αλλά μπορώ να σας απαντήσω πουθενά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ δεν φταίμε εμείς το κείμενο της Κομισιόν, το οποίο σας υπευλήθη, το οποίο θα το τροπολογήσετε και θα συναποφασίσετε με το Συμβούλιο. Δεν το έχει. Τώρα, τι είναι μια χορτολιβαδική έκταση μόνιμη, αν θέλετε. Το καθορίσαμε εμείς αυτό. Δεν κάναμε τον ορισμό. Όταν μιλάμε για διατήρηση αυτού του είδους των εκτάσεων, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο, πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το επίπεδο. Σήμερα δεν το ξέρουμε. Ποια, πόσες χιλιάδες εκτάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται ως μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις. Τι πρέπει να μετά το 2020. Ούτε εμείς το ξέρουμε, την Κομισιόν ούτε εσείς. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα λοιπόν. Υπάρχει μία ασυνέπεια στους στόχους. Επίσης, ο ορισμός εγώ ως μέλος της, του ελεγκτικού συνεδρίου δεν είμαι η Δήμων, ούτε αρμόδιος να πω κάτι τέτοιο. Αλλά η έννοια αυτή, το μόνο το οποίο κάνει, είναι να γίνεται όλο και πιο σημαντική όταν συζητούμε. Και σήμερα τι μπορούμε να πούμε, ότι ένα δάσος επειδή προσφέρει δέντρα που σκιάζουν την περιοχή γύρω είναι χορτολιβαδική έκταση. Για να δώσω μόνο έναν ορισμό, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα δώσω εγώ τον ορισμό αυτό. Και μία παρατήρηση για το εισόδημα. Να απαντήσει την κυρία Μαγκίνος που έθεσε το θέμα αυτό ιδιαίτερος. Στην παρέμβασή μου, και αυτό δεν είναι καινούριο, το, έχω πει, το έχουμε πει και το έχουμε γράψει διάφορες εκθέσεις. Διαπιστώσαμε ότι η ΚΑΠ γενικά συνεισέφερε ουσιαστικά στο υποστήριξη των εισοδημάτων των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. σε Ανατολή και Δύση. Παρακαλώ. Νομίζω ότι καλό ήταν το συμπέρασμα αυτό στο οποίο καταλήξατε, δεδομένου ότι πρέπει σύντομα να αποχωρήσουν οι διερμηνείς και νομίζω ότι καλά ήταν αυτά τα τελευταία λόγια που είπατε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Χρειαζόμαστε διάλογο, χρειαζόμαστε κάποιες έννοιες, κάποιους ορισμούς να τους κάνουμε πιο ακριβείς. Σας ευχαριστώ και πιστεύω ότι αυτή η κοινή συζήτηση μεταξύ μας μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Αύριο, όπως είπαμε, στις 10 προβλέπεται η συνάντηση των συντονιστών και η Επιτροπή μας θα συνεδριάσει από τις 11. Ευχαριστώ και συγγνώμη που στο τέλος σας έκανα να βιαστείτε λίγο. Αλλά ήταν ενδιαφέρουσα η συνάντηση, ακούσαμε διαφορετικές απόψεις και αποκλίνουσες. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας.